We are starting the meeting. I would like to welcome everybody and open the, this first meeting of the AFCO committee after. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στη συνεδρία Επιτροπής μας μετά από τις διακοπές. Η συνεδρίαση αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο. Το πρώτο θέμα είναι η υιοθέτηση φυσικά της ημερήσιας διάταξης. Σας απεστάλλει στις 27 Αυγούστου. Έχουμε κάποιες αλλαγές εδώ. Γιατί ο Παύλο Ρανχέλ στο σημείο 8 για την έκθεση της ΕΚΟΝ για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών αναβάλλεται. Θα ήθελα να σας προτείνω ή απαιτείται κάποια πειθαρχία, να γίνει η απαιτείται κάποια πειθαρχία να γίνει η ψηφοφορία για τις δύο προτάσεις αμέσως μετά τις ανακοινώσεις, να είστε έτοιμοι να ψηφίσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση. Συνεπώς λοιπόν <clears throat> θεωρείται δεκτή η ημερήσια διάταξη εφόσον δεν υπάρχουν διαφωνίες. Δεν βλέπω κάποιο. Στο σημείο 2 να σας ανακοινώσω ότι θα υπάρξει μια έκτακτη συνεδρίαση την 28η Σεπτεμβρίου το απόγευμα. Αυτό γιατί θέλουμε να προετοιμαστούμε για την ψηφοφορία της Δευτέρας Οκτωβρίου στην Ολομέλεια για τον Ευρωπαϊκό Εκλογικό Νόμο. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι πριν το τέλος του Σεπτέμβρη. Θα έχουμε επίσης και μία συνάντηση με τον Φερχόστατ που θα μας ενημερώσει. Ελπίζω να καταφέρει να έλθει και να μιλήσει. Οι ανακοινώσεις οι σχετικές με τις ανακοινώσεις των συντονιστών ε, θα τις πω αργότερα για να μην σας καθυστερήσω. Πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων του μηνός Μαΐου. Είναι διαθέσιμα και θα θεωρηθούν δεκτά εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση πριν το τέλος αυτής της συνεδρίασης. Περνάω στο 6 και στο 7 τώρα γρήγορα, ψηφοφορίες. Θα ήθελα ξεκινώντας να δώσω το λόγο ή μάλλον στον Ρίτζαρ Κόμπετ, ναι, για την ερμηνεία του ε, του άρθρου 130. Έχετε μπροστά σας το κείμενο το οποίο συμφωνήθηκε στην ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση του κανονισμού ομόφωνα. Έχουμε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις μπροστά μας. Δεν θέλω να ξεκινήσει εκ νέου η συζήτηση επί της ουσίας αλλά από την τελευταία αυτή συνεδρίαση κάποιες πολιτικές ομάδες θεώρησαν ότι είναι λίγο ακραία η ερμηνεία αυτή, ιδιαίτερα το δεύτερο τμήμα της, ε, ότι δεν αρκούμεθα στην ερμηνεία των κανόνων ως έχουν, αλλά προσθέτουμε σε αυτούς. Ε, διαβουλεύτηκα λοιπόν με τους συντονιστές των ομάδων που μου είπαν ότι είχαν κάποιες δυσκολίες και γι' αυτό έκανα μία πρόταση να διαγράψουμε το δεύτερο τμήμα της ερμηνείας αυτής και η ερμηνεία του κανόνα του συγκεκριμένου, του άρθρου του συγκεκριμένου να περιοριστεί στις δύο πρώτες φράσεις. Να ερμηνεύσουμε αυστηρά δηλαδή ε, μέσω εξαιρέσεων, της φράσης μέσω εξαιρέσεων ή μέσω αποκλήσεων. Και δεν μπορεί οι εξαιρέσεις να είναι περισσότερες από ό,τι ο κανόνας. Όταν ο κανόνας λέει 5 δεν μπορεί κανείς συστηματικά να λέει 6 λόγω ακριβώς της ρύθμισης αυτής. Και γι' αυτό λοιπόν απορρίπτουμε το δεύτερο τμήμα. Και αυτό μπορεί να γίνει δεκτό από ό,τι κατάλαβα από όλες τις πολιτικές ομάδες ή τουλάχιστον έτσι κατάλαβα. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να σχολιάσει κάτι. Για το 191 δεν υπάρχει κάτι εδώ. Μπορούμε παρακαλώ να ψηφίσουμε. ανατάσσεως των χειρών. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ της ερμηνείας του 130, ποιος είναι κατά, αποχή, δεκτό. Και ερμηνεία τώρα του 191, ποιοι είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Δεν απέχει κανείς δεκτό. Έχουμε τους δύο εμπειρογνώμονες μαζί μας. Yeah, so I, So I'd like to, to move to point five on our agenda, which is the... Uh, Σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, συζήτηση για την επαναδιαπραγμάτευση της συνταγματικής σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι συνέπειες ε, αυτής της διαδικασίας θα ήθελα επί τη ευκαιρία σε δύο λεπτά να κάνω μια εισαγωγή στη συζήτηση. Πολύ εξημών ε, στην αίθουσα αυτή, αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξουν νέες μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα υπάρξουν, θα υπάρξουν μεταρρυθμίσεις ειδικότερα στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, ε, ε, σημαντικές μεταρρυθμίσεις και συμφωνούμε ότι σε περιπτώσεις κρίσεων, όπως για παράδειγμα κρίσεις ε, σαν τη μεταναστευτική κρίση ή την κρίση με τη Ρωσία και άλλου είδους κρίσεις, θα μας οδηγήσουν ενδεχομένως σε νέους τομείς ευρωπαϊκής πολιτικής και θα εμβαθύνει ε, το ρόλο της ε, ευρωπαϊκής δράσης. Παράλληλα βλέπουμε ότι η πολιτική ελίτ η Βρετανική λαμβάνοντας υπόψη αυτή την ε, μελλοντική προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ε, θέλουν να ε, προκαλέσουν τον αντιταχθεί η κοινωνία της Μεγάλης Βρετανίας την Ευρώπη της όλο και μεγαλύτερης συνεργασίας. Ο David Κάμερον εδώ και πάρα πολύ καιρό προσπαθεί να επιτύχει το να παραμείνει μέσω αναθεωρημένων ε, όρων ε, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν αυτά τα τέσσερα καλάθια που αναφέρει και το έγγραφο. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι η άποψη των ε, κρατών μελών από τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο σε σχέση με τις βρετανικές προσδοκίες. Είναι δύσκολο για μας σήμερα να το κρίνουμε αυτό. Αυτό επίσης που μας προκαλεί έκπληξη είναι ότι η βρετανική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει επισκέψεις ε, αλλά και ε, αναθεώρηση της δυνατότητας ε, ανακατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι επαρκές κάτι τέτοιο και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα χρειαστεί επαναπατρισμός σε επίπεδο συνθήκων, αλλά είναι γεγονός ότι πολλά στοιχεία παραγνωρίζονται στη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς, ωστόσο, θα θέλαμε να τονίσουμε ε, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θεωρούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της, πολιτικές ε, ε, οι οποίες υπέστησαν τεράστιες και εις βάθος ε, μεταρρυθμίσεις κατά τα τελευταία χρόνια και κατά τις τελευταίες δεκαετίες και μάλιστα υπό την επιρροή του Ηνωμένου Βασιλείου. Οπότε για μας είναι μάλλον παράδοξο να ακούμε πολιτικές ελίτ να αναφέρουν το ακριβές αντίθετο. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Ε, καταλαβαίνω ότι θα υπάρξουν πολλές συζητήσεις ε, ε, κατά, τα επόμενα, κατά τους επόμενους μήνες ότι το θέμα αυτό θα έχει όλο και περισσότερη πολιτική σημασία. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άκουσε τον Γκίφερ Χόφσταντ εχθές, τον πρόεδρο των Φιλελευθέρων και προσκάλεσε και τον Ντέιβιτ Κάμερον στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Πιστεύουμε ότι χωρίς τη σημερινή συζήτηση ε, με τους ανθρώπους που είναι οι πλέον οι δήμονες σε αυτό το θέμα, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πραγματική συζήτηση και να συμμετέχουμε και εμείς στη συζήτηση που λαμβάνει η χώρα. Τρεις εμπειρογνώμονες, δυστυχώς ο ένας ε, ε, ο καθηγητής Δεβίτες δεν μπορούσε να έρθει, όμως είναι εδώ ο Charles Grant, ο οποίος ε, ε, επί πολλά χρόνια ήταν επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κέντρου, είναι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού ε, Κέντρου Μεταρρυθμίσεων και ήταν πολύ συχνά παρόν εδώ στην κεντρική Ευρώπη και ο Ζων Κλοντ Πυρίς, τον οποίο δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά τουλάχιστον εδώ και 20 χρόνια ε, είστε εδώ γύρω και είστε επίσης ε, η ήσασταν επισκεφαλής ε, του, της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υπάρχουν λοιπόν, είναι εδώ παρόντες άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση. Ελπίζουμε ότι θα είναι επικοδομητική συζήτηση και μόλις μαθαίνω ότι ο Γκί Φερχόφστατ θα ήθελε να μιλήσει λίγο πριν από τους εμπειρογνώμονες γιατί πρέπει να φύγει. Να σας δώσω λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και κυρίως την Επιτροπή Συνταγματικών ε, Θεμάτων που οργάνωσε αυτή την συζήτηση. Μόνο να επαναλάβω αυτά που είπατε μπορώ, ότι σήμερα το πρωί η διάσκεψη των Προέδρων έλαβε την απόφαση να προσκαλέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον David Cameron. Ο κύριος Σούλτς ε, σήμερα το απόγευμα θα έρθει σε επαφή με την Downing Street για να δει ε, πώς ακριβώς θα γίνει αυτό. Αν δεχθεί την πρόσκληση αυτή, πώς θα οργανωθεί η επίσκεψή του και τι μορφή θα λάβει αυτή η ε, συνεδρίαση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για τα, τα αιτήματα της ε, Μεγάλης Βρετανίας δεν μπορούν να γίνουν και κλεισμένων των θυρών. Πρέπει να είναι διαφανής ο τρόπος συζήτησης και ο καλύτερος τρόπος είναι η πρόσκληση του Βρετανού Πρωθυπουργού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν αυτό οργανωθεί, τότε η Επιτροπή, η σας πρέπει να παίξει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, δεν ξέρω ακριβώς πώς, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ενημερωθείτε ε, κατά πόσο ο Πρωθυπουργό θα αποδεχθεί αυτήν την πρόσκληση και πώς θα την οργανώσουμε. Τούτου λεχθέντος, ε, το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να θέσω, είναι το Ε, Επειδή έχω δύο φορές κάνει φωτοσχόλιο στην ΑΦΚΟ για την έκθεση την οποία επεξεργαζόμαστε με τον ε, κύριο Μπρόκ και την κυρία Μπρεσό πέρα από τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι ένα από τα βασικά ζητήματα της έκθεσης. Πόσα opt-out μπορεί κανείς να έχει και να εξακολουθεί να αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό ζήτημα ε, και τώρα ε, έχουμε και όλα αυτά τα αιτήματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι δύσκολο, καταλαβαίνουμε βέβαια ότι υπάρχουν ε, εξελίξεις, ίσως κάποιοι να μπορούν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό, αλλά το πρώτο είναι να καταλάβουμε ποιες ε, ποια είναι τα αιτήματα αυτά της Μεγάλης Βρετανίας και γι' αυτό ακριβώς ε, η διάσκεψη των Προέδρων θεώρησε ότι ήταν απολύτως αναγκαίο να προσκληθεί ο Πρωθυπουργό ε, David Cameron για να ακούσει ακριβώς ποιες είναι οι απαιτήσει της Βρετανικής πλευράς. Μία τελευταία παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία ε, των εργαζομένων. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Το όλο θέμα αυτό συνδέεται με την κρίση τη μεταναστευτική που βιώνουμε στην Ευρώπη. Έτσι έχουμε δημιουργήσει κατά κάποιο τρόπο ένα καζάνι που όλα βράζουν μέσα Ίσως πρέπει να είναι λίγο σαφέστερος ο ορισμός της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα να ενισχύσει το δικό του εθνικό σύστημα για να αποφύγει πολλά προβλήματα και η κρίση των προσφύγων και των μεταναστών ε, και την κρίση των προσφύγων και των μεταναστών σήμερα γιατί είναι σαν να λέμε ότι τα δύο αυτά πράγματα είναι το ίδιο που δεν ισχύει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα δεν έχει καμία σχέση με το άλλο. Αυτό λοιπόν το οποίο εμένα με ανησύχησε πολύ είναι αυτό που μόλις σας ανέφερα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο κύριος Ποιής είναι εδώ. Με πολύ μεγάλη χαρά θα ακούσω τι έχει να μας πει. Πάντοτε ήταν συμμετείχε στις συζητήσεις ε, στο Συμβούλιο και θα ήθελα να ακούσω τη δική του άποψη για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ για να μην καθυστερήσουμε. Τέλος, είσαι ο πρώτος που θα μιλήσει στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ντανούτα. Το σύντομο έγγραφο που έχω το... έχει διανεμηθεί θα το διαβάσω γιατί θα πάρει πολύ χρόνο. Θα κάνω μόνο κάποια προκαταρκτικά σχόλια και στη συνέχεια θα αναφερθώ στα 10 προβλήματα, στους 10 παράγοντες που μπορεί να σημαίνει ότι αυτοί που είναι από τη δικιά μου πλευρά θα χάσουν το δημοψήφισμα. Αν ε, καταφέρει να πετύχει μια συμφωνία, ε, ο Κάμερον θα είναι μια πολύ μετριοπαθή ε, συμφωνία, δεν θα μεταμορφώσει τον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα υπάρχουν opt-outs για τη Μεγάλη Βρετανία. Θα παρουσιαστούν ω μεταρρυθμίσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίω και ίσω για ένα-δύο στοιχεία που αφορούν τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά δεν θα υπάρχουν πολλά opt-out. Το πρόβλημα είναι ότι ο Κάμερον θα πρέπει να το ε, παρουσίασαν ε, μια ε, μεταμορφωτική ενέργεια για να έχει την υποστήριξη για το δημοψήφισμα. Και αυτή θα είναι μια δυσκολία που θα αντιμετωπίσουμε εμεί οι προευρωπαϊστέ. Και υπάρχει και περίπτωση ο Κάμερον να δω, θέλει να θέλει να δώσει μια παραστατική μορφή στην τρόπο λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, όσον αφορά τα... τις παροχές προς τους ε, μετανάστες και τα λοιπά, είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι μόνο ε, οι αμόρφοι που υποστηρίζουν το UKIP. Οι πρόσφατες αστυγές δείχνουν ε, Ε, ότι υπάρχει μετανάστευση πάνω από 600.000 ε, υπάρχουν πάνω από 600.000 μετανάστες και το πρόβλημα είναι ότι η μετανάστευση σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές ε, χρησιμοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες και αυτό που έχει στην καμπάνια του ως πρόσχημα ο Νάιντερ Φαράζη λέει ότι ο μόνο τρόπο να κρατήσουμε την στην ε, Μεγάλη Βρετανία είναι να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, ο Κάμερον πρέπει να καταφέρει κάτι μέσα από όλα αυτά. Είπε βέβαια ότι θα προσπαθήσει να κάνει κάτι για τι ε, παροχέ υπηρεσιών για τα επιδόματα εντό τη εργασία. είναι όντως προβληματικό σημαντικό αυτό γιατί είναι, θα υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε άτομα από άλλα κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με την εισαγωγή του Universal Credit που θα είναι αυτό η μεταρρύθμιση στα, στην πολιτική των ρυθμάτων και αν αυτό ισχύει για όλους το απαραίτητο θα είναι κάποιο να ζήσει στο ΕΕ για κάποια χρόνια πρωτού ε, λάβει αυτό το επίδομα, τότε αυτό ενδεχομένω θα είναι νομικά εφικτό. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να πετύχει κάτι σε αυτό το πνεύμα και να σεβαστεί βέβαια το, την αρχή τη ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτό που θα αποφασίσουν θα επηρεάσει φυσικά τον αριθμό μεταναστών που θα εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί οι περισσότεροι έρχονται περισσότερο για να εργαστούν και όχι για τα επιδόματα. Ελπίζω οι κανόνες να γίνουν πιο δίκαιοι, να υπάρχει λιγότερη κατάξυση του συστήματος, ότι θα υπάρχει ένα πιο δίκαιο σύστημα που δεν θα ε, δημιουργεί μειονεκτήματα για αυτούς τους πολίτες που πληρώνουν τους φόρους τους κτλ. Ε, πιστεύω ότι και ο Ζαν Κλόντ θα έχει κάτι να πει από αυτού και ένα άλλο θα μου πούνε πολύ σημαντικό είναι η σχέση ανάμεσα στα in και τα out. Αυτό δεν είναι θέμα για την κοινή γνώμη, αλλά πιο πολύ για τι επιχειρήσει για τους κυβερνητικού για τον όσπον, τον Υπουργό ε, Οικονομικών και για πολλού άλλου. Καθώς ολοκληρώνεται η Ευρωζώνη, ενδεχομένω να αρχίσει να λαμβάνει αποφάσει αποφάσεις ε, για μεγάλα ευρωπαϊκά θέματα που θα επηρεάζουν τα συμφέροντα της ενιαίας αγοράς. Never, but the recent example uh, just before the summer holiday of... Πριν τις δικοπές ε, του καλοκαιριού και την κρίσιμη σύνοδο για την Ελλάδα, αποφασίστηκαν να χρησιμοποιήσουν το EFSM για να δοθεί ένα δάνειο γέφυρα στην Ελλάδα, παρόλο που η ε, μεγαλύτερη ήταν ενάντια στη χρήση αυτό, μπόρεσαν και το περάσανε τελικά και έτσι ε, δημιουργήθηκαν ανησυχίες ε, στην ε, Βρετανική πλευρά. Επίσης, οι Γερμανοί θεωρούν ότι αυτό που θέλουν να πετύχουν οι είναι ένα βέτο για την πόλη του Λονδίνου μπορεί να το πιστεύουν αυτό οι Γερμανοί μετά το φιάσκο του 2000, του 2011. Θεωρώ λοιπόν ότι θα είναι δύσκολο να πετύχουμε μια συμφωνία γιατί οι Γερμανοί δεν έχουν δείξει συμπάθεια όμως ενδεχομένως κάτι να μπορεί να γίνει, να υπάρξει μια συμφωνία για ένα μελλοντικό άρθρο ότι τίποτα από αυτά που θα περάσει δεν θα βλάπτει την ε, εσωτερική αγορά. Και μια άλλη ιδέα που συζητιέται είναι να υπάρχει ένα είδος μηχανισμού ε, φρεναρίσματος κατά κάποιο τρόπο, όχι βέτο ακριβώς, αν μια, μια, ε, μια χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πει ε, ότι η Ευρωζώνη βλάπτει τα συμφέροντα της στήριξης αγοράς, να μπορεί ε, μια χώρα της Ευρωζώνης να χρησιμοποιήσει αυτό το μηχανισμό. Να πω τέλος κάτι για τα προβλήματα και το λόγο που θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο να πάρουμε να έχουμε αποτέλεσμα φαίνεται ναι. Ένα είναι η εσωτερική δυναμική του Συντηρητικού κόμματο, οι ευρωσκεπτικιστέ. Έχουν μάθει ότι αν πιέσουν τον Πρωθυπουργό και τον απειλήσουν να βιαστεί, πολλέ φορές αυτός υποχωρεί. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε τώρα το δημοψήφισμα, γιατί αρχικά ο Κάμερον δεν ήθελε να προτείνει δημοψήφισμα. Και φτάνουμε στο σημείο που ο Κάμερον πλέον δεν μπορεί να κρατήσει ικανοποιημένους τους ευρωσκεπτικιστές. Θα πρέπει σύντομα να έχει ένα πολύ, μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση στη, στα αιτήματά τους. Δεν θα μπορέσει να κάνει τις ε, ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις που θέλουν αυτοί είναι ο επαναπατρισμός και γι' αυτό θα του ζητήσουν ε, να κάνει ε, περισσότερα πράγματα. Έχουμε δει τον Μπόρις Τζόνσον τελευταία να λέει ότι θέλουμε να ανακτήσουμε το κοινωνικό opt-out που, που εισήγαγε ο Τζον Μέτζορ το 1991. Αν θέλει να κερδίσει λοιπόν το δημοψήφισμα, δεν θα μπορεί να βγάλει ένα λαγό από το καπέλο στη μαγεία στο τέλος. Είμαι αισιόδοξο, όμως θεωρώ ότι η εσωτερική δυναμική του Συντηρητικού κόμματο θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η ζημιά στο βρετανικό μπραντ. Το γεγονός ε, ότι η Βρετανία δεν θα δεχτεί πρόσφυγες που, από αυτούς που φτάνουν στην Ουγγαρία και στην Ιταλία και στην Ελλάδα δεν είναι και πολύ καλό για την εικόνα της Μεγάλης Βρετανίας. Ε, φαινόμαστε αντιπαθητικοί. Όπως είπε ο κ. Φερχόφστατ, το θέμα των, προσφύγων δεν είναι δύο με τις μετανάστευσεις. Τα έχουν κάπως ε, μπλέξει μεταξύ τους. Και έτσι παρουσιάζονται στα μέσα μας και ενημέρωσης. Ο ε, ε, ένας ε, υπουργό είπε ότι θα πρέπει να δεχτούμε 10.000 μετανάστε ε, στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά το κοινό πιστεύει ότι πρέπει να προσφέρουμε κάτι περισσότερο και έτσι δημιουργείται μια εικόνα που δεν είναι και τόσο συμπαθητική. Κατά τρίτον, και μιλώντα γενικά, πολλά άλλα κράτη-μέλη και θεσμικά οργάνα δεν θα θέλουν να αποδείξουν του Άγγλου γιατί το βρετανικό μπράντ δεν είναι και τόσο δημοφιλές. Αλλά πολλοί φοβούνται και τι επιλογέ που θα έχει ένα Brexit. Όποιε μεταρρυθμίσει και αν ε, αποφασιστούν ε, στο πακέτο του Κάμερον θα πρέπει να περάσουν από δυναμωτική οδό και να έρθουν και στο Ευρωκοινοβούλιο. ώστε να μειωθούν π.χ. τα επιδόματα στους ε, μετανάστες, ε, τη μείωση της γραφειοκρατίας κλπ. Ε, αυτά μπορεί να μην βρουν απήχηση και πολλές κυβερνήσεις επίσης δεν θα είναι και πολύ ικανοποιημένε με όλα αυτά. Κανείς δεν θα είναι πρόθυμος να υποχωρήσει τόσο πολύ ώστε να βοηθήσει τους Βρετανούς. Και αν υπάρχει κι άλλο ρεύμα μεταναστών από το της Μάχης, το χάρη, ένα μεγάλος, ένας μεγάλος όγκος ε, μεταναστών, τότε αυτό θα δημιουργήσει και άλλη πίεση. Επίσης, η κρίση της Ευρωζώνης, πάντα όταν υπάρχει μια σύνδοση κορυφή, υπάρχουν ε, αντιπαρθέσεις ανάμεσα στους ε, Γερμανούς και τους Έλληνες και έτσι οι Βρετανοί έχουν την εικόνα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα κακό χάλι. Και αυτό τους κάνει να ρωτιούνται αν θέλουν να παραμένουν προσκολλημένοι σε ένα οικονομικό πτώμα. Αλλά όσο αναζωπηρώνεται αυτή η κρίση, τόσο πιο πολλοί οι συμπολίτε του πατριώτε μου θεωρούν ότι δεν είναι και τόσο καλό ε, να είμαστε συνδεμένοι με αυτέ τι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλο, ανησυχώ για την εκστρατεία για να μείνει η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μια ε, εξαιτία από τα πάνω προς τα κάτω, δηλαδή Goldman Sachs και ε, διάφοροι θα προσπαθούν να υποστηρίξουν αυτή την εκστρατεία και θεωρώ ότι αυτό ότι θα, ε, αποτύχει γιατί η αντίθετη καμπάνια για την ε, έξοδο θα είναι από κάτω προς τα πάνω, θα είναι απλοί άνθρωποι που θα υποστηρίζουν όλα αυτά. Και το έβδομο σημείο, εξαιτία υπέρ του όχι, έχει πολύ ισχυρά επιχειρήματα. Αν αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά θα μπορούμε να συνεχίσουμε τι εμπορικέ σχέσει. Η Κίνα δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχει εμπορικέ συναλλαγέ. Δεν δεν θα υπάρχει ζημιά στι εξαγωγέ μα. Αν φύγει από το Ευρωπαϊκή Ένωση η Βρετανία, ε, τότε θα, οι να θα στα χέρια του λαού και θα μπορούν να, διαθέτουν κάποια κονδύλια για ε, π.χ. το σύστημα υγείας ε, στην ε, Μεγάλη Βρετανία, σε εθνικό επίπεδο δηλαδή. Και το 8ο σημείο είναι ότι η εργατική βρίσκονται σε μια κατάσταση αναταραχή. από το 1980 το εργατικό κόμμα είναι ένα κόμμα υπέρ της Ευρώπης και αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει τον τελευταίο χρόνο εξαιτίας των γεγονότων στην Ελλάδα την αντίληψη ότι ο Σόιμπλε έχει κάνει πολύ κακό στους Έλληνες ότι ε, μεταχειρίστηκαν άδικα το ΣΥΡΙΖΑ και το Τζίπρα και υπάρχουν και άλλοι λόγοι βέβαια. Αλλά στο Εργατικό Κόμμα έχουμε τον Τζέρμι Κόρμπεν και αυτοί που τον υποστηρίζουν ε, δεν τους ενδιαφέρει πιο πολύ η εξουσία αλλά θέλουν να είναι ηθικά στη σωστή πλευρά και ο Κόρμπαν ε, είναι αμφιλεγόμενος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ακριβώς εναντίον της αλλά θα βοηθήσει την εκστρατεία γιατί στο εργατικό κόμμα θα υπάρχουν εσωτερικές ε, αντιπαραθέσεις, ενδεχομένως διχασμός. Η περισσότερη είναι υπέρ της ε, Ευρώπης, ε, αλλά παρόλο ότι υπάρχει ακόμα πρόβλημα και το ένα το σημείο, το ένα το θέμα που υπάρχει, ο Ζακ Ντιλόρ και η Μάρκερ Θάτσερ ε, μας ότι είναι καλό πράγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ντελόρ γιατί έδωσε την κοινωνική διάσταση και υπήρχαν πολλά ωφέλη όπως ε, η αντιμετρότητα και άλλα τέτοια. η αρχηγοί των συνδικάτων μπορεί να υποστήριξουν το όχι, μπορεί και τον ένα ανάλογα με το τι θα του υποσχεθεί ο Κάμερον. Αλλά πιστεύω ότι ο Κάμερον δεν θα προσπαθήσει ε, να επαναπατρίσει πολλά από την κοινο... στον κοινωνικό τομέα, να επαναπατρίσει πολλούς. Και μετά έχουμε και τον επιστημικό κλάδο. Θυμάμαι το δημοσίευμα του 75, ήμουν 16 χρονών τότε, όλοι οι επιχειρηματίες μίλησαν υπέρ της παραμονής στην Ευρώπη. Αυτό δεν θα συμβεί πάλι τώρα, γιατί οι περισσότερε μεγάλε επιχειρήσει θέλουν να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πολλοί απλώ θα σιωπήσουν γιατί θα φοβηθούν ε, ε, να δημιουργήσουν ε, θέματα σε, στα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη, σε εμπορικού εταίρου κτλ. Οπότε οι περισσότερε επιχειρήσει πιστεύω ότι δεν θα εκφραστούν και τόσο έντονα. Και υπάρχουν και κάποιε επιχειρήσει που είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν του αρέσουν κάποιοι κανονισμοί. Υπάρχουν οι αμέτρες και σήμερα. Τότε ο Harold Βίλσον αποφάσισε να κάνει το νομοψήφισμα για να κρατήσει ενωμένο το εργατικό κόμμα. Πήγε στις Βρυξέλλες, επαναδιαπραγματεύτηκε και γύρισε με ένα χαρτί που έλεγε έχουμε μια καλύτερη συμφωνία για την Βρετανία. Προσπίθηκε ότι ήταν μια καλύτερη συμφωνία και τον πίστεψαν. Ο λαός τον πίστεψε γιατί έτσι το προβάλλαν τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό που έχει αλλάξει από τότε είναι ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα έχουν διαφορετική προσέγγιση, διαφοροποιημένη προσέγγιση. Θα το σκηθεί πολύ μεγάλος έλεγχος Κάμερον από το κόμμα του και από τους άλλους. Άρα δεν θα είναι εύκολο να κερδιθεί το δημοψήφισμα και αν θεσμικά όργανα όπως εσείς μπορείτε να βοηθήσετε περνώντας κάποιους νόμους, αυτό θα ήταν χρήσιμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Jean-Claude Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Έχει περάσει λίγος καιρός και βεβαίως θα διαφωνήσω με τον Κίφερ Χότστατ. και θα πω ότι δεν εκπροσωπώ, τη... δεν εκπροσωπώ το Συμβούλιο. Ξέρετε ότι έχω φύγει εδώ και πολύ καιρό ε, και μόνο προσωπικές απόψεις ε, θα εκφράσω σήμερα. Συμφωνώ με την ε, εικόνα που παρουσίασε ο Charles Grant και για, τα, για τους διάφορους κινδύνους που υπάρχουν με το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Όμως αυτό δεν είναι λόγος να μην είμαστε διορατικοί για το τι μπορούμε να κάνουμε ή τι μπορούμε να αποδεχθούμε όταν θα παρουσιάσει το Ηνωμένο Βασίλειο τις απόψεις του. Καταρχάς, θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος. Φανταστείτε τι θα μπορούσε ο κύριος Κάμερον ε, να διαλέξει ως στρατηγική για τις διαπραγματεύσεις, ποιος θα είναι ο βασικός στόχος των διαπραγματεύσεων αυτών. Υπάρχουν διάφορα σημεία αφετηρίας και οι πιθανότητες επιτυχίας τους κατά την άποψή, μας, ε, την άποψή μου είναι πολύ διαφορετικές. Σύμφωνα και βέβαια και για τη συνταγματική ε, θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι διαφορετικό να λέει κανείς τι θα γίνει σε περίπτωση που παραμείνει η ε, Μεγάλη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαφορετική τι θα γίνει σε περίπτωση Brexit. Το θέμα της αναθεώρησης τώρα των συνθήκων ε, σύμφωνα με την άποψη του καθηγητή Ντεουί, ο οποίο απέστειλε ε, στην ΑΦΚΟ το, την εισήγησή του, το καθεστώς θα μπορούσε να διατηρήσει την ε, Μεγάλη Βρετανία ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν μέρη όμως δεν θα συμμετέχει σε άλλες ε, ε, πολιτικές ή θα επιλέξει να συμμετέχει ή να μη συμμετέχει σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, στην κοινωνική πολιτική, στην εξωτερική πολιτική κλπ. Να κάνω καταρχάς ένα σχόλιο όσον αφορά την ε, πολιτική. Το χρονοδιάγραμμα. Η ιδέα είναι να προταθεί η αποδοχή ενός νέου καθεστώτος ε, στο, για το Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς είναι δυνατόν να κάνει κανείς δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να μην ξέρει την απάντηση των υπολείπων χωρών. Αν ε, γίνει πρώτα το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι αδύνατο κάτι τέτοιο γιατί δεν ξέρει κανείς οι, τα 27 κοινοβούλια ή τα 25 δημοψηφίσματα που μπορεί, τα 27 δημοψηφίσματα που μπορεί να γίνουν. Ε, κάποια θέλουν δημοψήφισμα, κάποια κράτη-μέλη ε, ζητούν απλώς ε, κοινοβουλευτική έγκριση. Ξέρετε λοιπόν ότι τώρα οι ηγέτες των ευρωπαϊκών ε, κρατών δεν θέλουν μια τέτοιου είδους ανοιχτή συνθήκη και να ε, ε, υπάρξουν συγκεκριμένες συνθήκες που θα αφορούν απλώς τα εσωτερικά ζητήματα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι θα είναι δυνατόν να δρομολογήσει κανείς αυτή τη διαδικασία πρώτα στα κράτη-μέλη, χωρίς να ξέρει κανείς κατά πόσο ο Βρετανικός λαός θα το αποδεχθεί αυτό και να γίνει αυτό κάτι τέτοιο σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ε, το να πάει κανείς ε, πρώτα στο Βρετανικό λαό και να ρωτήσει, χωρίς να γνωρίζουν εκείνοι ποια είναι, ποια είναι η άποψη των υπολείπων κρατών μελών, και αυτό είναι αβέβαιο. Τι γίνεται λοιπόν τώρα με την περίπτωση του πρώτου σεναρίου ένα τέτοιο είδους αίτημα ε, για το ειδικό καθεστώς ε, θα ήταν τόσο θεμελιώδους ε, σημασίας από συνταγματική απόψης, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι τα υπόλοιπα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να δεχθούν μια τέτοιου είδους αρχιτεκτονική, η οποία ουσιαστικά είναι μια επιλογή διάλεξε και πάρε για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί θα αλλάξει θεμελιωδώς ε, της αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αυτονομία της αν ένα κράτος μέλος ή ένα εν μέρη μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις ε, αποφάσεις της Ένωσης και αν γίνει αποδεκτό στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα ανοίξει την πόρτα και για άλλες χώρες όπως Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία ή ακόμη και ε, από μέλη της Ένωσης. Αυτό το σενάριο λοιπόν είναι πραγματικά ε, εντελώς απίθανο να επιτύχει. Δεύτερο σενάριο που είναι ο επαναπατρισμός των ε, εξουσιών, των αρμοδιοτήτων που ανέφερε ο Τσάρλς. Αν γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να ισχύσει για όλους βάσει της συνθήκης και έχω και το, τις ίδιες παρατηρήσεις για το χρονοδιάγραμμα που είχα και για το πρώτο σενάριο. Από πολιτικής απόψεως ε, δεν είναι ρεαλιστικό. Τα ζητήματα που έχουν αναφερθεί ε, άπτονται σημαντικών και βασικών αρχών όπως η κυκλοφορία των πολιτών, ε, η ισότητα μεταξύ των ε, διαφόρων κρατικών θεσμών και ζητήματα όπως το κοινωνικά κεφάλαια ή τα διαρθρωτικά ταμεία. Και επί της ουσίας βέβαια είναι ε, δεν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Ακόμη και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ε, είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει οργανώσει μια μεγάλη έκθεση τριών χιλιάδων σελίδων. Το αποτέλεσμα, το συμπέρασμα της οποίας λέει ότι μια κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποδεκτή. Τρίτο σενάριο. Το τρίτο σενάριο είναι το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει στην Ένωση ως μέλος όμως θα γίνουν αλλαγές στη συνθήκη που ή θα ε, σημαίνει ότι θα είναι πιο ακριβή η συνθήκη σε κάποιες πτυχές, κάτι που θα ισχύει για όλα τα κρατη ή να, έχει ακόμη περισσότερα opt-outs, συγκεκριμένα το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα μπορούσε κανείς, βάσει των ετοιμάτων που υποθέτουμε ότι θα καταθέσει το Λονδίνο και αναφέρθηκε και ο Τσάρλς σε αυτή την πιθανότητα, Όσον αφορά το Ever Closer Union, δηλαδή την ένωση όλο και μεγαλύτερη συνεργασία, ε, συγκέντρωση της εξουσία στα εθνικά κοινοβούλια και έλεγχο της επικουρικότητας ε, ε, της, και της νομοθεσίας βάσει αυτής τη αρχής της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη δυνατότητα μετακίνησης κυκλοφορίας ενός πολίτη από το ένα κράτος μέλο τη Ένωση στο άλλο. Θα υπάρξει λοιπόν μία αλλαγή της συνθήκης. Το πρώτο ερώτημα το πρώτο θέμα είναι ότι υπήρξε κάποια παρανόηση σε σχέση με την, ε, ε, με, την νομική ερμηνεία ότι υπήρξαν δηλαδή κάποιες παρανοήσεις και παρεξηγήσεις ε, σε σχέση με το τι θα πει Ευρωπαϊκή Ένωση ολοένα και μεγαλύτερη συνεργασία. Δεύτερον, υπάρχει το θέμα της Ευρωζώνης που θα συνεχίσει να υφίσταται στο μέλλον. Ε, όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, πρέπει να ληφθούν υπόψη δυνατότητες μεγαλύτερης νομικής προστασίας για τα κράτη-μέλη που είναι εκτός Ευρωζώνης και τα κράτη-μέλη, ε, κατά τρίτον, χρειάζονται τη βοήθεια των εθνικών κοινοβουλίων για να γίνεται σεβαστή καλύτερα αρχή της επικουρικότητας που είναι μια πολιτική έννοια και όχι νομική έννοια και τη βελτίωση της δημοκρατικής νομιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα τρία λοιπόν πρώτα θέματα. Εγώ δεν διαφορώ με το να αλλάξουμε, δεν με το να αλλάξουμε κάποτε τη συνθήκη. Το τέταρτο όμως μου δημιουργεί πρόβλημα γιατί αφορά ένα συνταγματικό ζήτημα βασικό που είναι η ισότητα μεταξύ των πολιτών. Τώρα, για τα τρία πρώτα ε, θέματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να επιτύχει ένα τέτοιο σενάριο αυτή τη στιγμή, κατά την τρέχουσα περίοδο, ακόμη και για αυτά τα τρία, ε, για αυτές τις τρεις περιπτώσεις. Γιατί κάθε απόπειρα αλλαγή της συνθήκης, ε, δικαίως κατά τη γνώμη μου, θα ανοίγει τη συζήτηση για την αναγκαιότητα βελτίωση, βελτίωσης της δημοσιονομικής βάσης της Ευρωζώνης. Και επειδή η πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο το να ανοίξει αυτός ο πολύ σημαντικός φάκελος που κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει. Οποιαδήποτε αναθεώρηση των συνθήκων κατά πάσα πιθανότητα ε, λόγω της ε, συγκυρίας θα απορριφθεί. Μερικά ακόμη θέματα, ε, μερικά σχόλια ακόμα για ε, αυτά που είπε ο Charles Grant στην εισήγησή του. Το να έχει κανείς ε, την ίδια πολιτική άποψη για το θέμα αυτό όπως η δική μου και λέει εκείνος στην εισήγησή του ότι μπορεί αυτό το εμπόδιο να ε, το αντιπαρέλθουμε άμα γίνει αν γίνουν κάποιες αλλαγές ε, στη συνθήκη. Είναι κάτι που έγραφε και ένα άρθρο της Financial Times. Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα είναι όμως λόγια. Πρόκειται για μια πολιτική δήλωση πρόθεσης, το οποίο δεν δεσμεύει τα, τις αποφάσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων και υπάρχει και μια ακόμη πρόταση από τον Steve Pierce ε, που έχει δημοσιευθεί, και προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ε, μετατρέποντας την υπόσχεση σε κάτι το νομικά δεσμευτικό. Το πρόβλημα με αυτή την ιδέα είναι ακριβώς ότι το να γίνει νομικά δεσμευτική μία υπόσχεση και να ε, μεταγραφεί σε συνθήκη θα παραβιάζει το άρθρο 48 της ε, ε συνθήκης που λέει ότι δεν είναι δυνατόν να αλλάζει η συνθήκη κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί κανείς ε, να ε, αλλάξει κάτι, έστω και με μια νομικά δεσμευτική τέλος πάντων υπόσχεση, να αλλάξει κάτι τέτοιο ε, την ίδια την ε, ε, συνθήκη της Ένωσης. Γι' αυτό οι αποφάσεις 209 και 1992 δεν συμπεριλαμβάνουν τέτοιου είδους υποσχέσεις απλώς διευκρινίζουν τις υφιστάμενες ε, διατάξεις της συνθήκης και είναι, ε, συνάδουν 100% με τη συνθήκη. Και έχει επιβεβαιωθεί και με, με ε, απόφαση, την απόφαση Ρότμαν του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2010. Αν λοιπόν προσθέσει κανείς κάτι ή αν την σημασία της συνθήκης, δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό ακριβώς εγώ πιστεύω ότι αυτές οι υποσχέσεις δεν είναι ε, κάτι το πάρα πολύ καλό, εκτός εάν ε, το Ηνωμένο Βασίλειο δεχθεί ε, δήλωση προθέσεων που δεν έχουν καμία νομική ισχύ. Τέταρτο και τελευταίο σενάριο που είναι το εξή. Το Ηνωμένο Βασίλειο, με λίγη βοήθεια βέβαια των φίλων του, να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την αλλαγή των συνθήκων. Αλλά πολιτικά μέτρα να υπάρξουν και αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις των ε, λειτουργιών και των μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αναγνωρίζοντας ε, το γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των προβλημάτων που ανέφερε και ο Τσάρλς και συμφωνώ, είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς, μου φαίνεται ότι κατά τη γνώμη μου είναι το πιο υποσχόμενο και το πιο ρεαλιστικό σενάριο θα υπάρξουν κάποιες, θα γίνουν κάποιες ε, ε, μεταρρυθμίσεις που ζητάει ο Κάμερον αποδεκτές, αλλά πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες άλλων ε, κρατών θα ήθελαν τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις σαν αυτές που ζητάει ο Βρετανός Πρωθυπουργός και νέα πολιτικά μέτρα. Για παράδειγμα, ένα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ε, της ε, εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών συγκεκριμένα, δρομολόγηση της ε, εθελοντική συνεργασίας πολιτικών ενέργειας και διαφόρων άλλων τομέων, βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών των ευρωπαϊκών και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να αρχίσουμε από τη δήλωση του 2014 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να υπάρξει ένα επίσημο κείμενο με αυτή τη βάση κάτι το οποίο θα διασκεδάσει τις ε, λαμφασμένες ε, ερμηνείες ε, και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, θα έλεγα ότι πρακτικούς τρόπους για τη μείωση της γραφειοκρατίας, για τη βελτίωση του σεβασμού της επικουρικότητας, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων και τέταρτον, που είναι και το πιο δύσκολο, όπως είπε ο Τσάρλς, για την καλύτερη προστασία των ε, ε, ε, μελών των πολιτών της Ένωσης και η σχέση μεταξύ των χωρών εντός και εκτός Ευρωζώνης είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ευπρόσδεκτο στο πλαίσιο αυτό. Θα μου πείτε τι γίνεται με το πέμπτο σενάριο που είναι το Brexit, η έξοδος της ε, Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ξέρετε ότι μπορεί να συμβεί και κάτι τέτοιο. Σίγουρα η Βρετανική κυβέρνηση έχει εξετάσει εις βάθος το ενδεχόμενο αυτό και έχει συνειδητοποιήσει ότι κάτι τέτοιο θα είναι αρνητικό για τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ένα Brexit θα μπορούσε να σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι δορυφόρο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, γιατί θα βρίσκεται στην κατηγορία της Νορβηγίας, της Ελβετία κλπ. ή θα είναι εντελώς απομονωμένο μόνο του και πρέπει από την αρχή να επικυρώσει όλες τις εμπορικέ συμφωνίες, όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με τι υπόλοιπε χώρε του κόσμου, ενώ η διαπραγματευτική δύναμη ε, που θα έχει δεν θα είναι πια τόσο σημαντική, ούτε είναι τόσο σημαντική όσο πιστεύουν ορισμένοι. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, αναλαμβάνω, πρώτον, δεν θα πρέπει να αποτελεί ταμπού κάτι τέτοιο η αναθεώρηση των συνθήκων. Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο και μπορεί να γίνει. Όμως, μία αλλαγή ε, της συνθήκης από πολιτικής ε, απόψης είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ε, για τους λόγους που εξήγησα προηγουμένως, ε, γιατί υπάρχει και το θέμα της ενίσχυσης της Ευρωζώνης. Η τρέχουσα πολιτική συγκυρία δεν θα ε, συμφωνούσε με μια σύντομη λύση βραχυπρόθεσμη, κάτι το οποίο χρειάζεται στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεύτερον, δεν είναι δυνατόν πια η Ευρωπαϊκή Ένωση με 28 ετερογενείς χώρες να επιμείνει σε μία ε, λύση. Πρέπει λοιπόν να αποδεχθούμε το γεγονός ότι υπάρχει μία ασύμετρη, ε, μια πιθανότητα ασύμετρης ολοκλή, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο μέλλον, θα υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία και ότι αυτό δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη τις επιθυμίες όλων των κρατών μελών και δεν κολυσιεργεί. Υπάρχουν όμως και ε, θεσμικά όρια τα οποία πρέπει να σκεφτούμε. Και ο Τσάρλ συμφωνεί μαζί μου. Πρώτον θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις από την πολλαπλή αυτή γεωμετρία όπως η ενιαία αγορά, ο ανταγωνισμός και λοιπά Δεύτερον, θα πρέπει να διατηρήσουμε την αυτονομία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτούς τους τομείς. Τρίτες χώρες μπορεί να ωφελούνται από την ενιαία αγορά, αλλά δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θα πρέπει να διατηρήσουμε λοιπόν τα βασικά χαρακτηριστικά του κοινοτικού δικαίου, δηλαδή κυριαρχία του κοινοτικού δικαίου, ενιαία ερμηνεία. Και τέλος θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εν την πλήρη αυτών σύνθεση εφόσον υπάρχουν μορφές ε, ε, ενισχυμένης συνεργασίας για τις οποίες είναι υπεύθυνα και θα πρέπει επίσης να υπάρξει απόλυτο σεβασμό της ενίας πράξης. Τα όρια αυτά θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο σεβασμού σε όλες τις περιπτώσεις και από το Ηνωμένο Βασίλειο. Συνταγματικά λοιπόν, αν αποσυρθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο θα περιπέσει στην κατάσταση της Ελβετίας και της Νορβηγίας θα γίνει ένα είδος δορυφόρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να υιοθετήσει νέα μέτρα σχετικά με τα κενά της ε, ε, εσωτερικής αγοράς. Και αν αρνηθεί ε, να σεβαστεί τους κανόνες αυτούς, τότε θα πρέπει να διακόψει τους δεσμούς με την ενιαία αγορά και να διαπραγματευτεί εκ του μηδενός. Όπως είπε και ο κ. Φερχώστατ προηγουμένως, αυτά είναι τα βασικά συνταγματικά προβλήματα γύρω από την περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας. Σόλτς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο μιλητές για τις ε, ενδιαφέρουσες αναλύσεις τους για ένα πολύ περίπλοκο θέμα. Όταν συζητήσαμε το θέμα αυτό στο παρελθόν, είχα κάνει μια παρατήρηση. Ένας πολίτης με ρώτησε τι γίνεται με την παρούσα κρίση στον τομέα το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Ρώτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρηθεί, θα διασωθεί ή θα αναγκαστεί να κλείσει ουσιαστικά λόγω αυτών των κυμάτων των μεταναστευτικών. Θα πρέπει λοιπόν με σοβαρό τρόπο να προσπαθήσουμε να δούμε τι είναι η μεταναστευτική πολιτική και τι συνέπειες έχει για το μέλλον και το θεσμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, βασιζόμενο στις παρατηρήσεις σας, is Μήπως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει κάτι περισσότερο από μία απλή ενιαία αγορά, από έναν απλό χώρο αγοράς έτσι ώστε οι λαοί που συναποτελούν την Ένωση να βρουν πραγματικά ε, ένα ενδιαφέρον στα πλαίσια αυτής της δομής. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνδέεται με τις συζητήσεις, τις πολιτικές και τις οικονομικές γύρω από την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά όχι μόνο. βλέπει κανείς ε, τα ερωτηματικά που θέτουν οι πολιτικές δυνάμεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι απαντήσεις δίδουν στις ερωτήσεις τις οποίες θέτουμε. Και μπορούμε να θέσουμε το θέμα αυτό και στις δικές μας χώρες σε επίπεδο συνταγματικό γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να χάνουμε το χρόνο μας με τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου, εφόσον οι πολίτες πολλές φορές δεν γνωρίζουν γιατί ψηφίζουν. Είναι ένα από τα ερωτήματα λοιπόν. και σαν συνέπεια αυτής της προβληματικής θα πρέπει να οργανώσουμε κάποιες συζητήσεις τώρα και να δώσουμε απαντήσεις. Σε επίπεδο όμως πολιτικής, η πολιτική πρόκληση είναι να καταφέρουμε να δώσουμε στους πολίτες της Ένωσης ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τις θέσεις μας, τις πολιτικές μας θέσεις, τις θέσεις των πολιτικών μας κομμάτων. και έτσι θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε και τα μέσα για να ανταποκριθούμε στις επερχόμενες συνέπειες προβλημάτων όπως αυτό. Θα πάρουμε ερωτήσεις και μετά θα ζητήσουμε από τους δύο μιλητές να αντιδράσουν. Σεφλίν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δύο μιλητές για τις ενδιαφέρουσες αναλύσεις σας. οι ερωτήσεις μου προς τον Τσάρλ, αλλά φυσικά και προς τον επόμενο μιλητή. Αυτό το οποίο δεν γίνεται δεκτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει το Ηνωμένο Βασίλειο σε επίπεδο δημοψηφίσματος. Αναφερθήκατε κι εσείς στην αύξηση του αριστερού ευρωσκεπτικισμού και στο εργατικό κόμμα. Υπάρχει δυνατότητα διέρεσης του εργατικού κόμματος γύρω από το δημοψήφισμα. Η δυναμική αυτή θα οδηγήσει σε διάσπαση του εργατικού κόμματος. Δεύτερη ερώτηση. Τι αντίληψη επικρατεί στη Μεγάλη Βρετανία για τους δύο εκατομμύρια Βρετανούς που ζουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Τρίτο σημείο. Δεν αναφερθήκατε στη Σκοτία. Θα ήθελα τη γνώμη σας για τη Σκοτία. Εσείς θα δώσετε τις απαντήσεις, καταλαβαίνετε όμως τι εννοώ. Όταν μιλήσατε για τις λεγόμενες αντικαθεστοτικές εκστρατείες, εγώ είχα πάρει μέρος σε εκστρατείες στο παρελθόν. Αλλά τώρα τι γίνεται ακριβώς με τα μέσα δικτύωσης, τα κοινωνικά μέσα. Ε, θα κινητοποιήσουν τους πολίτες, θα κινητοποιηθούν τα μέσα αυτά. Γιατί έχουν μεγαλύτερο ρόλο να παίξουν από τα τελευταία δέκα χρόνια. Πάντα μου κάνει εντύπωση η πάρα πολύ σκληρή αντιευρωπαϊκή γραμμή, διεστραμμένα σκληρή μερικές φορές, στα λαϊκά μέσα ενημέρωσης τι ακριβώς θα συμβεί ε, με, την, ε, με τα υπόλοιπα μέσα, με την τηλεόραση και με τις ε, σοβαρές σε εισαγωγικά εφημερίδες, τα μεγάλα φύλλα. Εδώ φαίνεται να υπάρχει ένα παράδοξο. Από τη μία φαίνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνεί σε σχέση με την Ευρωζώνη με κάποιες από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Από την άλλη όμως στον τομέα της μετανάστευσης υπάρχει μια πλήρης διάσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν αναφέρομαι σε χώρες οι οποίες είναι pre-in, δηλαδή έτοιμες να μπουν, αλλά αναφέρομαι και σε χώρες όπως η Λιθουανία, η Ουγγαρία που είναι μέλη. Ευχαριστώ, Τζόρτζ. Λάινεν. Ευχαριστώ πολύ. Τα συμπεράσματά σας ε, συμφωνούν. Πολιτικές δηλώσεις, πολιτικές αναλήψεις υποχρεώσεων για μεταρρυθμίσεις μελλοντικέ. Απαιτείται περισσότερη καθαρότητα, περισσότερη ευκρίνεια. Για να αλλάξουμε την Ένωση πρέπει να αλλάξουμε τις συνθήκες και να αποκτήσει καινούριο χαρακτήρα η Ένωση. Εγώ νομίζω ότι το δημοψήφισμα είναι κάτι το ιδιαίτερα επικίνδυνο. Έχουμε εμπειρίες ε, για δημοψηφίσματα για την Ευρώπη, η οποία δεν είναι πολύ κοντά στις ανησυχίες των πολιτών και δεν απαντά στα προβλήματα των πολιτών, αλλά δείχνει να τους θέτει προβλήματα. Θα συμφωνήσω λοιπόν μαζί σας ότι τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται μέχρι τώρα είναι απλουστευτικά. Και υπάρχει χώρος έτσι ώστε να οικοδομηθεί μια αποτελεσματική φιλοευρωπαϊκή εκστρατεία. Μήπως όμως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές στα ερωτήματα τα οποία τίθενται. Το πρώτο ερώτημα είναι αν θα παραμείνει η Ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η, το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα το ερώτημα τίθεται με διαφορετικό τρόπο. Θα μείνουμε ή θα φύγουμε. Η διατύπωση είναι διαφορετική και ο τρόπος με τον οποίο τίθεται μια ερώτηση την κάνει λιγότερο ή περισσότερο επικίνδυνη. Τσάρλς είπε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου ο Κάμερον θα έχει βάλει στη σειρά τα μέλη του κόμματός του. Αλλά τι θα γίνει αν μέλη της κυβέρνησης του εκστρατεύσουν υπέρ του όχι. Θυμάστε το δημοψήφισμα για το ευρώ πριν μερικά χρόνια και ο Υπουργός Οικονομίας ήταν κατά του ευρώ. Αν λοιπόν η ίδια η κυβέρνηση δεν είναι ενωμένη, τότε πώς μπορεί να περιμένει κανείς νέα αντίδραση από το λαό. Για να μην μακρηγορήσω, θα συμφωνήσω ότι οι βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να φυγούν. Όχι πλέον opt-out, όχι πλέον αποκλήσεις εξαιρέσεις, Έχουν πάρα πολλές εξαιρέσεις ήδη ορισμένες χώρες. που δημιουργούν ειδικέ συνθήκες, υποτίθεται καλύτερες συνθήκες για το Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι το οποίο είναι εναντίον του πνεύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέτει σε αμφισβήτηση την ισότητα των κρατών μελών. Αν τυχόν συνεχίσουμε με τη λογική του να βρούμε ειδικέ καλύτερε συνθήκε για κάθε χώρα ξεχωριστά, τότε να το κλείσουμε το μαγαζί. Μεγαλύτερη λοιπόν εναρμόνιση και όχι μεγαλύτερες εξαιρέσεις. Ε, οι ατομικές ελευθερίες είναι κόκκινη γραμμή. Η κοινοτική μέθοδος είναι κόκκινη γραμμή. Μπορεί και δεν υπάρχει βέβαια ακόμα το σύστημα της κόκκινης κάρτας, όπως και της πράσινης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βλέπουμε πως δουλεύει η ΚΟΖΑΚ. Το Westminster, η Γερουσία η Γαλλική και η Γερουσία η Ολλανδική θέλουν να υπάρξει ε, μια δυνατότητα αρνητικής αντίδρασης μέσω της ε, κίτρινης κάρτας ήδη. και αντιδρούν με τον τρόπο αυτό αντί να τους δίνουν κόκκινη κάρτα επειδή παρεμβαίνουν ε, στην κοινοτική μέθοδο. Σίγουρα να γίνει πιο ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό επιδιώκουμε και με την ε, βελτιωμένη ε, νομοθετική δραστηριότητα. Πρέπει να δούμε τι Ευρώπη θέλουμε. Μια απλή Ευρώπη ελευθέρου εμπορίου. Θέλουμε όμως και προστασία των δικαιωμάτων, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία των καταναλωτών. Ο ανταγωνισμός δεν είναι τα πάντα. Αν συγκεντρώσουμε μόνο την προσοχή μας στον ανταγωνισμό, μιλάμε για άλλη Ευρώπη. Λοιπόν, ελπίζω αυτό το οποίο παίζει ο Κάμερο να μην είναι ρωσική ρουλέτα, να μην στραφεί το Ηνωμένο Βασίλειο εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να μην χρησιμοποιηθεί η διαφορά αυτή για εσωτερικούς ε, λογαριασμούς, ξεκαθάρισμα εσωτερικών λογαριασμών στο εργατικό κόμμα. ο Κόρμπετ και στη συνέχεια οι συνάδελφοι θα απαντήσουν. Νόμιζα ότι είμαι ο μόνος Βρετανός προβουλευτής που μιλάει σε αυτό το διάλογο. Να πω πρώτα ότι εγκρίνω την, απόφαση της διάσκεψης των Πρόεδρων να καλέσουν τον David Cameron. Είναι κάτι που πραγματικά αξίζει. Αλλά όσον αφορά αυτά που ακούσαμε από τους ε, Δύο μιλωτέ, τα δέκα πράγματα που μπορούν να πάνε στραβά, αυτά που ανέφερε ο Τσάρλ στην παρουσίασή του, θα πρέπει να μα ε, κάνουν να ανησυχήσουμε. Υπάρχουν πράγματι πολλά πράγματα που μπορούν να πάνε στραβά, χωρί πρόθεση και να συμβεί ε, ένα Brexit ω ατύχημα. Δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Και υπάρχει και η τρέλα, που, ε, η τρέλα του να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία που οφείλεται εν μέρη στους ε, διαφορές που υπήρχαν μέσα στο συντηρητικό κόμμα. Η ε, μία από τα δεν θέλει να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό οποιασδήποτε συνθήκε και η πιο μετροπαθή πτέρυγα θεωρεί ότι όλα αυτά είναι τρελά. Ειδικά αυτοί που είναι κοντά στι επιχειρήσει και υπάρχουν και διάφορες αποχρώσεις στο ενδιάμεσο. Και για να κρατηθεί αυτό το κόμμα ενωμένο πριν τι εκλογέ, ο Κάμερον είπε ότι μετά τι εκλογέ, θα διαπραγματευτούμε ρυθμίσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια θα αφήσουμε του πολίτε του Μηνοβασιλείου να αποφασίσουν, χωρί να σκεφτεί καν ότι θα χρειαστεί όντω να φέρει αποτελέσματα, αλλά θα μπορούσε να τα διαπραγματευτεί στο πλαίσιο μια κυβέρνηση ανασπισμού μετά τι εκλογέ. Γιατί ούτε στην ίδια περιμέναν ότι θα κερδίσουν την απόλυτη πλειοψηφία και τώρα είναι παγιδευμένοι γιατί κάνουν την υπόσχεση και τώρα θα πρέπει να την τηρήσουν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως, είναι να παρουσιάσουν μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια διαδικασία που είναι διαρκής. Αυτό κάνουμε εδώ συνεχώς. Αναθεωρούμε ευρωπαϊκές πολιτικές ε, και νομοθεσίες οι περισσότερες νομοθεσίες που ψηφίζουμε εδώ είναι ουσιαστικά τροποποίηση προηγούμενων νόμων. Αυτό κάνουμε λοιπόν και εμείς και το Συμβούλιο, μεταρρυθμίσεις και αναθεωρήσεις. Υπάρχουν πολλές μεταρρυθμίσεις ε, καθοδόν. που θα μπορούσαν να τις χρησιμοποιήσουν ε, οι συντηρητικοί. Παραδείγματο χάρη το ReFit, ε, ο οργανισμό για την ε, για better regulation, είναι η κοινή ελευθερική πολιτική. Μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλά που συμβαίνουν και που είναι προ όφελο όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει αυτό ο Πρωθυπουργό και να πει ναι, αυτά του χρειαζόμαστε. Αλλά Αντιθέτως τι έκανε. Έκανε μια δικά, δικιά του, έκανε δικό του κατάλογο ασκώντας πιέσει στο κόμμα του. Στην ομιλία του Bloomberg, ε, στο Bloomberg που πρότεινε το δημοψήφισμα δεν έκανε λόγο για τη μεταρρύθμιση ε, στη, μεταναστευτικό ε, στο θέμα των μεταναστών που εισέρχονται στη Μεγάλη Βρετανία και για ποιο λόγο γιατί εντωμεταξύ είχε δεχτεί πιέσει από τη δεξιά πτέρυγα του κόμματο που θέλανε ε, που του έθεσαν ε, τεράστιες απαιτήσεις γιατί θέλανε ουσιαστικά να αποτύχει. Άρα κινείται κάπου ανάμεσα σε λεπτομέρειες που δεν είναι τόσο σημαντικές κάτι στο οποίο θα είναι εύκολο διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχει από την άλλη πλευρά και αξιώσει, οι οποίε όμω είναι αδύνατο να τι πετύχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα κινείται ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα. Θα πρέπει να βρει κάτι ώστε να βοηθήσει στο δημοψήφισμα και να το κερδίσει. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως. Αν είχα πιο πολύ χρόνο, θα αναφερόμουν σε όλα αυτά που είπε προηγουμένως ο Τσάρλς. Μιλάμε για μια όλο και πιο ενωμένη ένωση, όπως αναφέρεται στο ε, προήμιο της συνθήκης. Γίνεται, γίνεται λόγος και για την επικουρικότητα Κάτι που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευση και για τον Τζον Μέιτζορ. Όλα αυτά όμω δεν αλλάζουν κάτι. Είναι ε, λεπτομέρειε, είναι ασήμαντα. Αν μπορούν να το βοηθήσουν, καλώ. Αλλά ανάμεσα σε αυτά τα ασήμαντα και τα αδύνατα, τα διανόητα, θα πρέπει να βρει κάτι να κάνει, όπως πήγε ο κύριος Πύρης, με βοήθεια από τους φίλους του, γιατί δεν θα είναι εύκολο και κανένα από εμάς, από ό,τι φαίνεται. Ένα τελικό ερώτημα στον κύριο Πύρης. Αν υπάρξει αλλαγή στη συνθήκη, και αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι επιθυμητό και θα είναι και επίση πολύ δύσκολο, αλλά κάποια πράγματα από αυτά που θέλει ο Κάμερο δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω από δευτερεύουσα νομοθεσία γιατί θα, ε, θα πρέπει να παραιτηθούν στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και για αυτό το λόγο αν ο κύριος Κάμερο δεν απαιτήσει αλλαγή συνθήκης αλλά ένα πρωτόκολλο επί θα μπορεί να συμφωνηθεί ώστε να προσθεθεί στη συνθήκη για αυτό το χρόνο, μόνο στην επόμενη συνθήκη. Ένα τέτοιο σενάριο χρησιμοποιήθηκε για την Ιρλανδία και ξέρω κύριε Πύρες, είπατε ότι η Ιρλανδία δεν άλλαξε ε, τις θεμελιώδες αρχές ε, της συνθήκες, αλλά υπήρξε η υπόσχεση, η δέσμευση ότι θα εισαχθεί αυτό το πρωτόκολλο και θα προσθεθεί στη συνθήκη. Και το οποίο έγινε όταν προσχώρησε και η Κροατία. Θα μπορούσε να συμβεί κάτι παρόμοιο και σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, όλα ξέρετε το περιεχόμενο, αλλά από πολιτική πλευρά, θα μπορούσε αυτό να ήταν ένα ενδεχόμενο σενάριο που θα χρησιμοποιούσε η Βρετανική πλευρά. Θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω κάποιε ερωτήσει στον Ζαν Κλοντ Πύρη, ακριβώ σε δύο θέματα, το πρωτόκολλο Θυμάσαι την ε, ειδική πλειοψηφία και τη συνθήκη της Λισαβόνας και τι συνέβη τότε. Οπότε υπάρχουν δυνατότητες ενδεχομένω να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Και το δεύτερο ερώτημα που έχω να κάνω είναι αυτό που Δεν υπάρχει ε, διάθεση να αλλάξουμε τη συνθήκη. Γιατί δεν υπάρχει διάθεση από τα κράτη-μέλη. Αλλά τι πιστεύετε πρέπει να γίνει για να υπάρξει αυτή η διάθεση για την αλλαγή της συνθήκης. Τι πρέπει να συμβεί για να ουσιαστικά να αλλάξουν άποψη τα κάθε μέλη. Υπάρχει κάποιο βρετανικό όραμα για την Ευρώπη. Γνωρίζεις αν υπάρχει κάποια στοιχεία που να συνθέτουν αυτό το όραμα, με το οποίο θα ήταν ευχαριστημένοι οι Βρετανοί. Θα έχουμε ακόμα έναν ομιλητή, γιατί έχουμε πολύ μακρύ κατάλογο. Ο κύριο Τάσκ, είστε εδώ, ναι, ο λόγος εσάς. Jedno słowo najpierw. E, wydaje mi się, że więcej dobrego zrobimy, jeśli będzie. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι μπορούμε να κάνουμε θετικά πράγματα. Αν αναζητήσουμε δυνατότητες αντιμετώπιση των προβλημάτων με θετικό τρόπο. Νομίζω ότι αυτό είναι καλύτερο από το να περιοριστούμε στο να κατηγορούμε το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι παρουσιάσουν την άποψη ότι αντιμετωπίζουμε, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο σαν ασθενή, το οποίο έχει ανάγκη θεραπείας. Εγώ δεν θέλω να περιοριστώ στην κριτική, θέλω να βρω λύσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούει κανείς αυτά τα οποία θα μας πει ο κύριος Κάμερον, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε σε στενή επικοινωνία με την Επιτροπή και με το Συμβούλιο. Και εκεί ίσως να ακούσουμε και κάποιες διαφορετικές ιδέες από αυτές που ακούσαμε εδώ. Ο Αντιπρόεδρος Τίλεμανς είπε ότι θα ήταν διατεθειμένος να κάνει κάποιες διορθώσεις έτσι ώστε να αποφευθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ η ιδέα αυτή του κυρίου Τίμερμανς δεν είναι μια ιδέα με την οποία είμαι σύμφωνος, αλλά παρόλα αυτά δείχνει ότι υπάρχουν επιμέρους στοιχεία διαπραγμάτευσης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω να παραμείνουμε σε επαφή με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Νομίζω ότι οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο θα είναι ομόφωνες αλλά ίσως όμως και όχι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικές. Θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις και στους δύο εμπειρογνώμονες συγκεκριμένες. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν οι Βρετανοί χωρίς αλλαγές στη συνθήκη σε τομείς όπως η ενίσχυση του ρόλου των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Και δεύτερον, θεωρείται ότι είναι δυνατόν να ξεπεραστούν τα προβλήματα και οι διαφορές στην ερμηνεία που υπάρχουν στον τομέα του εργατικού δικαίου. αλλαγές στη συνθήκη είναι απαραίτητες για να υπάρξουν επιμέρους αλλαγές ε, στις ε, νομικές ρυθμίσεις της κάθε χώρας. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. Κύριο Πύρης, ευχαριστώ. Για το πιο σημαντικό για μένα θέμα που είμαι δικηγόρος συμφωνία ενός πρωτοκόλου για το μέλλον. Ο κύριος Πίρς, καθηγητής Πίρς, έχει γράψει γι' αυτό. Δυστυχώς αυτός είναι λάθος τρόπος. Είναι λάθος τρόπος γιατί ποτέ στο παρελθόν δεν έχει υπάρξει η περίπτωση να υιοθετηθούν αποφάσεις αρχηγών κρατών, από πλευράς αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Μετά από το πρώτο αρνητικό δημοψήφισμα συνέβη με τη Δανία, με την Ιρλανδία και στις δύο περιπτώσεις οι αποφάσεις οι οποίες έγιναν δεκτές είναι απόλυτα σύμφωνες και σύμβατες με την ισχύουσα συνθήκη. Δεν υπάρχει ούτε ένα μικρό κόμμα το οποίο να διαφέρει. Το πρωτόκολλα αυτά δεν τροποποιούν τίποτα, δεν προσθέτουν τίποτα, απλά διασκρινίζουν. Στην ουσία δηλαδή είναι σαν ένα διακηρυκτικό κείμενο, τίποτα άλλο. Οπότε λοιπόν δεν θα πρέπει να έχετε την ψευδέστηση ότι μπορείτε να υιοθετήσετε μία απόφαση η οποία λέει ότι εφόσον προσθέσουμε κάποια πρωτόκολλα στη συνθήκη τότε θα έχουμε αλλάξει τη συνθήκη. Δεύτερον λέγω. Πρόεδρε εσείς ρωτήσατε το τι θα πρέπει να αλλάξει για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα το οποίο να οδηγήσει στις αλλαγές των συνθήκων. Νομίζω ότι η οικονομική ανάπτυξη θα βοηθήσει έτσι ώστε να βελτιωθεί το πολιτικό κλίμα και πολύ σημαντικό είναι επίσης να υπάρξει μια πίεση από πλευράς της πολιτικής ηγεσία. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια όθηση από πλευράς της πολιτικής ηγεσία και να δοθούν οι εξηγήσει τις οποίες περιμένει το κοινό. Το κλίμα όμως έτσι όπως είναι σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μια άλλη ερώτηση. Για το τι είναι εφικτό να γίνει κανείς έτσι ώστε να κερδίσει τις καρδιές των Βρετανών. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα λαμπρό και ευγενές, αλλά στο συγκεκριμένο αυτό δημοψήφισμα είναι εντελώ διαφορετικό από τα προηγούμενα. Στα προηγούμενα έπρεπε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει το τι υπάρχει μέσα σε μια τεράστια νέα συνθήκη, στη συνθήκη του Μάστρη. Κανένας δεν διάβαζε, κανένας δεν κατανοούσε, είναι περίπλοκα κείμενα. Αντίστοιχα και με τη Λισαβόνα, περίπλοκη κατάσταση, Έχετε τα αποτελέσματα των αρνητικών δημοψηφισμάτων στη Γαλλία και τις κάτω χώρες. Και βασικός ο λόγος ήταν γιατί ο κόσμος δεν καταλάβαινε. Τώρα όμως τα πράγματα είναι ανάποδα. Είναι εντελώς αντίθετη η κατάσταση. Αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν υπέρ της περιπέτειας, υπέρ του αγνώστου. Η Λισαβόνα και το Μάστριχτ ήταν λίγο περιπετειώδεις προτάσεις. Το ίδιο και τώρα δημιουργείται μια κατάσταση η οποία είναι κατάσταση που οδηγεί στο άγνωστο. Δεν ξέρουν αν θα είναι καλό για τα προσωπικά τους συμφέροντα και για τα συμφέροντα της χώρας τους να πούν όχι. Τώρα για τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν εδώ να αλλάξουν οι συνθήκες. Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε με πρακτικούς τρόπους τα κοινοβούλια των κρατών μελών να φέρουν εις πέρας καλύτερα τις αρμοδιότητές τους στα πλαίσια της επικουρικότητας και στα πλαίσια της Λισαβόνας. Να βοηθήσουμε τα κοινοβούλια να συντονιστούν, να βοηθήσουμε τα κοινοβούλια να αποκτήσουν περισσότερο χρονική, περισσότερη χρονική άνεση, γιατί έχουν πολύ λίγο χρόνο για να αντιδράσουν σε νομοθετικές προτάσεις. Και δεύτερον, να εμπλέξουμε περισσότερο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περιπτώσεις όπου γίνονται προτάσεις από αρκετά κοινοβούλια, από έναν δεδομένο αριθμό, η Επιτροπή θα πρέπει να το αντιμετωπίζει με σοβαρό τρόπο. Το ερώτημα που μου ετέθη είναι κατά πόσο οι Βρετανοί βλέπουν αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι τίποτε παραπάνω από μία αγορά η άποψη των Βρετανών είναι κάπως ανάμεικτη. Γιατί ναι, οι περισσότεροι Βρετανοί ως ε, ε, οικονομικό εγχείρημα το βλέπουν περισσότερο. Γι' αυτό ήθελα να μείνουν στο 1975. Αν, παραμείνουν, αν θελήσουν να παραμείνουν εντός της Ένωσης είναι γιατί φοβούνται τι θα γίνει από οικονομικής απόψεως αν φύγουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Ε, ε στην ε, Μεγάλη Βρετανία, όσον αφορά για παράδειγμα τις άδειες μητρότητας, πατρότητας, ε, ε, οι ώρες εργασίας κλπ. Είναι πράγματα τα οποία για τον απλό κόσμο δεν είναι πάρα πολύ δημοφιλή. Υπάρχει και το θέμα της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της αιρεσιμότητας και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μεταδώσει, έχει μεταδώσει την δημοκρατία, την ισότητα ισότητα σε ολόκληρη την Ήπειρο, ε, κάποια πράγματα τα καταλαβαίνουν, αλλά βασικά τη θεωρούν ένα οικονομικό εγχείρημα. Για την αριστερά με ρωτήσατε επίσης. Ένα πράγμα είναι να λέει κανείς ότι η αριστερά γίνεται, τάσεται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται πιο πολύ άκρα αριστερά και λιγότερο κέντρο αριστερά, για να, να σας το εξηγήσω έτσι. Και η ελληνική κρίση, Σόιμπλε, Ναντίον Τσίπρα, όλα αυτά είχαν τεράστιο αντίκτυπο ε, σε, στην ενίσχυση των απόψεων της αριστεράς, της άκρας αριστεράς, ε, γιατί φάνηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι ένα απλώς ένα μαστίγιο κατά των υπολείπων ο Ζων Κλοντ θα μπορούσε ίσως να μας εξηγήσει ε, κατά πόσο θα έχει και εκτιμένα δικαιώματα η Μεγάλη Βρετανία αν αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας το πούν αυτό οι νομικοί. Η Σκοτία βέβαια είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αν αποχωρήσει η Μεγάλη Βρετανία ε, από την Ένωση, η Σκοτία ε, θα έλεγε ότι θα ήθελε να παραμείνει, οπότε θα έπρεπε να γίνει, θα έπρεπε να, θα, θα να γίνει δεύτερο δημοψήφισμα για το αν θα παραμείνουν εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, οπότε θα, ψήφισαν θα, θα να βγουν. Ένα λοιπόν, μια παράπλευρη απώλεια θα ήταν η Σκοτία. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω τα προσόντα να σας μιλήσω για τα ε, κοινωνικά ε, και τη χρήση τους. Υποθέτω ότι δυστυχώς ε, ε, είναι ευρωσκεπτικιστικά περισσότερο από ότι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, τι να σας πω. Θα πρέπει να κάνουμε ένα σεμινάριο, μια μερίδα κάποια άλλη στιγμή για να σας το εξηγήσω αυτό. Εμέρη είναι η πώληση εφημερίδων το θέμα. Οι καλές, οι ωραίες ιστορίες, ε, συνήθως ε, οι ε, αντιευρωπαϊκές ιστορίες είναι πιο ε, διασκεδαστικό να τη διαβάζει κανείς από τις ιστορίες υπέρ της Ένωσης. Και γι' αυτό το όχι, για να το πω χοντρά, διαβάζεται περισσότερο από ότι το ναι ή οτιδήποτε είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει συνεχώς πίεση ε, από τους ευρωσκεπτικιστές ε, ε, στα μέσα ενημέρωσης που λένε στις εφημερίδες και στα, μέσα, τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης ότι είστε προκατηλημένοι, μεροληπτείτε υπέρ της Ένωσης κλπ. Οπότε υφίσταται τεράστια πίεση. Και αυτό έχει αλλάξει πολύ ειδικότερα μετά το 2004, όσον αφορά τη ρητορία για τη μετανάστευση ε, ναι, πράγματι έχει κοστίσει σε συμμάχους ε, στην ε, Μεγάλη Βρετανία. Ε, ίσως επειδή δεν έχουν α, οι, υπόλοιποι άνθρωποι που δεν ασχολούνται τόσο με το city ε, και τον αντίκτυπο που θα έχει μια έξοδος από το city, τους απασχολούν άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα οι μετανάστες. το ερώτημα, το, αυτό που είπε ο Τζο Λάινεν. Το νέο ερώτημα νομίζω ότι είναι καλύτερο από το, η νέα διατύπωση είναι καλύτερη από την πρώτη κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω ποια, θα πάρει, ποια απόφαση θα πάρει ο Κάμερον ε, για ε, την κυβέρνησή του. Ε, αν ας πούμε κάποιοι εγκαταλείψουν την εκστρατεία, ε, την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της εκστρατείας πριν από το δημοψήφισμα, δεν ξέρω τι απόφαση θα πάρει. η εργατική αν ο Κάμερον και ο Όσμπορν πρωτοστατήσουν και αν το ναι επικρατήσει, τότε μπορεί και άλλοι άνθρωποι όπως ο Βόρι Τζόνσον τελικά να αποφασίσουν να υποστηρίξουν ε, τον Κάμερον. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει. Τώρα για τα εθνικά κοινοβούλια που το έθεσε επίσης, συμφωνώ ε, με τον Ζων Κλοντ. Ξέρουμε τι θα γίνει. Θα υπάρξει μια ενισχυμένη διαδικασία κίτρινης κάρτας. Δεν θα είναι κόκκινη κάρτα. Όπως είπε ο Ζων Κλοντ, θα είναι πολύ πιο εύκολο οι εταίροι να συζητήσουν και να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Θα είναι δυσκολότερο για την Κομισιόν να πει όχι θα πρέπει να πάνε στο Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο ε, και να κάνουν ε, γύρω τραπέζι τρεις φορές αν υπάρχει μια κίτρινη κάρτα. Ρίτσαρτ Κόρμπετ. Α, αυτό θα το απαντήσει ο Ζων Κλοντ. Ντανούτα. Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σου. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει κανένα όραμα για την Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτοί που είναι υπέρ του όχι έχουν κάποιο ε, ο, όραμα. Ε, ο ε, βουλευτής του UKIP που έχει έτσι μια πιο προσγειωμένη θεώρηση σε σχέση με τον Φαράζ ε, θεωρεί ότι θα έπρεπε να είναι πολύ λιγότεροι κανόνες ε, ε, και θεωρεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα έπρεπε να είναι ένας πόλος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, έχει μια ιδέα και ο Τόνι Μπλερ είχε μια ιδέα σε σχέση με τη διεύρυνση, ήθελε να έχει μια ισχυρή εξωτερική πολιτική και γι' αυτό πρόθεσε τόσο πολύ την οικονομική μεταρρύθμιση και τη συνθήκη της Λισεβόνας. Και θα ήθελα να πω και κάτι θετικό. Αν και κερδίσουμε το δημοψήφισμα και θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, τότε πρέπει να ευχαριστήσουμε το κάμερο, τον Κάμερον, γιατί θα είναι η Μεγάλη Βρετανία ένα πολύ ευκολότερο σύμμαχος στο μέλλον, γιατί το λέω αυτό για την επόμενη γενεά πολιτικών. Ελπίζω ότι αυτό θα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα. Και το ε, τελευταίο ερώτημα, που αφορούσε και πάλι το το θέμα της κίτρινης κάρτας. Ε, η Βρετανική κυβέρνηση δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει με την πράσινη κάρτα. Εγώ συμφωνώ προσωπικά. Ναι, ε, τα εθνικά κοινοβούλια να υποβάλουν περισσότερες προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όχι. Employment law. Α, ναι, το εργατικό δίκαιο. μπορεί να, να υπάρξουν διακρίσεις. Για τα επιδόματα. Νομίζω ότι η απάντηση είναι όχι. Νομίζω ότι ο Κάμερον θα πρέπει να σεβαστεί τη βασική αρχή της ισότητας. Δεν μπορεί να ε, υπάρξουν τέτοιου είδους ε, ανισότητες. Ναι, για το τελευταίο συμφωνώ, λέει ο κύριος Πυρής για το ερώτημα που μου έθεσε ο Charles, αν υπάρχουν και κοιτημένα δικαιώματα για τους Ευρωπαίους πολίτες αν αποχωρήσει ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, το άρθρο 20 είναι κάπως αόριστο, αλλά συνδέει τα δικαιώματα ε, των πολιτών με την ιδιότητα του μέλους της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αν κάποιος Βρετανός υπήκος είναι σε μια άλλη χώρα, μέλος της Ένωσης, θα είναι σε λίγο διαφορετική θέση. Δεν θα έχει τα δικαιώματα ενός πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, βάσει της Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, θα διατηρήσουν την μόνιμη τους ε, ε, κατοικία αν έχουν μία. Για τους υπόλοιπους θα ισχύσουν, ε, θα το ισχύσει η τοπική νομοθεσία ε, ή ξέρω εγώ τα συμβόλαια, μια σύμβαση εργασία που του συνδέει. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα, όχι μόνο για του Βρετανού υπηκόου στι 27 υπόλοιπε χώρε, αλλά και για τι ε, υπηκόου των 27 χωρών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και είναι πολλοί αυτοί, όπω γνωρίζετε. Αυτό θα σήμαινε ότι θα υπάρξει ε, μία ε, διαπραγμάτευση και για το θέμα αυτό, αυτό να υπάρξουν ε, κάποια ειδικά μέτρα. Θα ήθελα να απαντήσω και στο Ρίτσαρντ, γιατί ρώτησε για το κείμενο της, όλο, της Ευρώπης όλο και περισσότερη συνεργασίας, Ever Closer Union. Ίσως θα ήταν καλό να υπάρχει ένα κείμενο ε, όχι νομικού χαρακτήρα, αλλά ήταν σημαντικό από πολιτικής απόψεως. Μια ε, γνωμοδότηση του δικαστηρίου και δεν είναι μόνο στο προήμιο, είναι και σε ένα άρθρο της ε, συνθήκης, όχι μόνο στο προήμιο. Είναι λοιπόν μια δέσμευση που δεν είναι ακριβής και αφορά τους λαούς της Ευρώπης, όχι τα κράτη, δεν... Όμως όλα αυτά πρέπει να υποθούν ε, γιατί το σεβασμό των ε, κρατών μελών, ε, το σεβασμό των συνδικών κλπ. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί υπήρξαν πάρα πολλές παρανοήσεις και παρεξηγήσεις στο βρετανικό τύπο. Θα είναι νομίζω πάρα πολύ χρήσιμο κάτι τέτοιο. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Στη Μάιτε τώρα λόγος. Είμαι Ισπανίδα και άκουσα όλα αυτά τα οποία είπατε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί είναι θέματα τα οποία πρέπει να παρακολουθήσουμε από κοντά. Μας ενδιαφέρουν όλους, μας αφορούν όλους. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά δείχνουν ένα μεγάλο επίπεδο αναξιοπιστίας ανευθυνότητας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να επηρεάσει το σύνολο φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως τη χώρα, το μέλλον της, την οικονομία της κτλ. Να σκεφτούμε λίγο τον Οδυσσέα. Τι θα είχε συμβεί αν ο Οδυσσέας στο ταξίδι του ανά τη Μεσόγειο, το τόσο περίπλοκο, είχε υποκύψει στα τραγούδια της Σιρήνας όταν ήταν δεμένος και δεν είχε δεθεί στο κατάρτι. Αν είχε υποκύψει από τις τις ειρήνες και θα είχε καταστραφεί. Δεν θα είχε φτάσει ποτέ στην Ιθάκη. Ποτέ δεν θα είχε ξαναδεί την οικογένειά του. Και fueran que hubiera tenido en su futuro sus proyectos, sus planes. Θα είχε αλλάξει τα σχέδιά του προφανώς. Λοιπόν, Ακούμε πάρα πολλά τραγούδια από τις σιρήνες, τις οποίες θα πρέπει όμως να μπορούμε να εντοπίσουμε. Θα πρέπει να δούμε τι μας τραγουδάει ο λαϊκισμός. Να δούμε φυσικά και τα λάθη τα οποία έχουν γίνει και ποιες είναι οι αδυναμίες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι τα τραγούδια αυτά από τις ειρήνες για να τα αποφύγουμε και να μην κάνουμε λάθη να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε οι μεν τους δε με μεγαλύτερη ευθύνη, με μεγαλύτερη υπευθυνότητα, να δούμε ποια είναι τα λάθη, έτσι ώστε να αποφύγουμε το λάθος και την καταστροφή της Ένωσης. πιστεύουμε ότι κάποιες από τις προτάσεις τις οποίες κάνουν οι Βρετανοί είναι προτάσεις οι οποίες αμφισβητούν τις βασικές αξίες των οργάνων μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι να αποφύγουμε τα τραγούδια αυτά. Είναι επικίνδυνες οι σιρήνες. Και όταν γνωρίζει κανείς τις λεπτομέρειες όπως εσείς γνωρίζετε στην ευρωπαϊκή πολιτική υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Και αν δεχτούμε κάποια πράγματα τα οποία φαίνονται ανώδυνα αυτό μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχει όμως ευθύνη βελτίωση των κοινοτικών οργάνων. Υπάρχει ευθύνη βελτίωση των κοινοτικών πολιτικών. Αλλά το βασικό πρόβλημα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε από κοινού και στα πλαίσια της αμοιβαίας κατανόησης. Και η ευθύνη εδώ κυρίως ε, πέφτει στα χέρια των Βρετανών ηγετών και της ε, Βρετανικής γενικά πολιτικής κοινής. Κάποια από τα πράγματα τα οποία μας είπατε ακούγονται καλά, αλλά μπορεί να κρύβουν παγίδες Eh, Mercedes Eh, grazie Presidente, eh, scuso anch'io parlerò. Θα μιλήσω την Ιταλική, λέει η Μπρέσο. Θα αντιστρέψω ε, το ερώτημα. Μήπως μπροστά στην ρεαλιστική υπόθεση την οποία έκανε λίγο πριν ο Κόρμπετ να υπάρξει δηλαδή ένα Brexit μη αναμενόμενο και να επηρεαστούν και οι υπόλοιπες 27 χώρες χώρες οι οποίες θα πρέπει να δώσουν μια απάντηση στα ερωτήματα, τα περίπλοκα τα οποία θέτει το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν έχουμε καταφέρει ε, να βρούμε μια λύση. Γιατί να μην αντιστρέψουμε λοιπόν το ερώτημα. Γιατί να μην πούμε ότι οι χώρες οι οποίες θέλουν μια πιο στενή μορφή συνεργασίας μια διαφορετική ένωση με μια κεντρική ιδέα πολιτική να αντιμετωπίσουν το θέμα της Ευρώπης των δύο ταχυτήτων. Και έτσι να δώσουμε την δυνατότητα στις χώρες που το επιθυμούν να μείνουν στο δεύτερο κύκλο, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε άλλες χώρες οι οποίες θέλουν να πάρουν μέρος μόνο στον εξωτερικό κύκλο. Αυτό θα επιτρέψει στις χώρες οι οποίες πρέπει να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις να μην τις κάνουν ουσιαστικά. Ή τουλάχιστον να μην το κάνουν τυχαία αλλά μέσω συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Όποιος θέλει να παραμείνει στον πυρήνα της, της πολιτικής Ευρώπης και όποιος θέλει μπορεί να παραμείνει στον δεύτερο κύκλο που είναι κυρίως η μορφή της οικονομικής συνεργασίας. Εγώ πριν λίγες μέρες πίστευα ότι αυτή θα μπορούσε να είναι μια λύση. Θα μπορούσε να παρουσιαστεί σαν μια λύση όχι μόνο για τη Μεγάλη Βρετανία, γιατί θα τεθεί πάλι εδώ ένα πρόβλημα, γιατί να δίδεται μια δυνατότητα τέτοια στη χώρα αυτή και όχι σε άλλες το πρόβλημα λοιπόν μιας διαρθρωμένης, μιας θεσμικής, οργανωμένης απάντησης, όχι τυχαίας, όχι περιπτωσιακής, είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο. Πριν λίγο καιρό έλεγα ότι αυτή η απάντηση θα ήταν μια σωστή απάντηση. Μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων μέσα στη συνθήκη. Εγκαταλείποντας κάποιες πιθανές αλλαγές για το μέλλον. Και έτσι να μπορέσουμε να προσφέρουμε λοιπόν στους σημερινούς και μελλοντικούς εταίρους την δυνατότητα να κάνουν την επιλογή τους. Το πρόβλημα όμως πριν λίγες μέρες, επίσημα νομίζω από την Υπουργό της Μεγάλης Βετανίας που ζήτησε να τεθούν περιορισμοί στην ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Εγώ είμαι στα πλαίσια της αντιπροσωπείας με την Ελβετία και είναι ένα θέμα που το έχουμε θέσει με ξεκάθαρο τρόπο σε μια χώρα που δεν είναι μέλος της Ένωσης. Αν θέλει κάποιος να παραμείνει μέσα σε μια ενιαία αγορά δεν μπορεί να αρνηθεί την ελεύθερη διακίνηση. Αν δεν υπάρχει ελεύθερη διακίνηση δεν υπάρχει Ένωση. Συνεπώς λοιπόν αυτό δεν μπορεί να ζητηθεί από μια χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλει ας φύγει, αλλά αν μείνει τότε θα πρέπει να δεχθεί ότι η ελεύθερη αγορά αφορά και την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα πάνω στο οποίο θα ήθελα την άποψή σας. Δεν βλέπω με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει την υπόθεση μιας επιμέρους ιδιότητας μέλους, μιας μερικής ιδιότητας μέλους. Αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε κατά περίπτωση να ορίζουμε το ποσοστό του ανήκει στην Ένωση. Αυτό είναι πάρα πολύ αδύνατο είναι να γίνει δεκτό συνολικά. Να έχουμε 18 ή 10-11 υποψηφιότητες σε διαφορετικό επίπεδο την κάθε μία. Αλλά για την ανιαία αγορά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένα κομμάτι της ενιαίας αγοράς αποτελείται από την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Και γι' αυτό δεν υπάρχει καμία διαφορά. Αυτό λοιπόν μου φαίνεται ότι είναι το πιο ευαίσθητο κομμάτι της συζήτησης. Και προς τα εκεί πηγαίνει η κατάσταση. Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό το θέμα από το θέμα των προσφύγων ή των παράνομων μεταναστών. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μια επίθεση από τη Βρετανική κυβέρνηση στους ίδιους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη Σκοτία ακούσαμε. θα φανεί ξεκάθαρο ότι η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας θα οδηγήσει και στην έξοδο της Σκοτίας. Αυτό βέβαια μπορεί να λειτουργήσει και αντίθετα. Μπορεί ίσως να κάνει τη Μεγάλη Βρετανία πιο διστακτική στο να κάνει αυτό το βήμα. Έχω πολλά να πω αλλά να μην σας κουράζω. Σας ευχαριστώ. Είναι πολύ χρήσιμες οι παρατηρήσεις σας. Porque me, Έχω την αίσθηση ότι το πλαίσιο στο οποίο προτείνονται οι συγκεκριμένες λύσεις δεν είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από τα αιτήματα τα οποία μας έχει θέσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι μόνον αυτό. Αυτό είναι μία κατεύθυνση την οποία παίρνει η συζήτηση. Υπάρχουν και άλλες κατευθύνσεις, υπάρχει και άλλη κατεύθυνση. Υπάρχουν πολλές ε, πολιτικές δυνάμεις, υπάρχουν πάρα πολλά πολιτικά επιχειρήματα υπέρ μιας Ευρώπης ισχυρότερης για να ξεπεράσει την κρίση. Μια Ευρώπη στην οποία πιστεύουμε πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα και της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και χριστιανοδημοκρατικά κόμματα που πιστεύουν και χρειάζονται μια Ευρώπη πιο ομοσπονδιακή. Μια Ευρώπη η οποία να έχει ισχυρότερο προϋπολογισμό σε σχέση με το 3 του ΑΕΠ. Μια Ευρώπη η οποία να είναι ε, περισσότερο ε, νομιμοποιημένη δημοκρατικά με ισχυρότερο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ένα ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονομικών που θα διαχειριστεί καλύτερα το χρέος της και την οικονομική της διακυβέρνηση. Υπάρχει λοιπόν στην Ευρώπη ένα πολιτικό ρεύμα πολύ σημαντικό που θέλει περισσότερη Ευρώπη. Εάν λοιπόν τώρα για να παραχωρήσουμε ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο την δυνατότητα να μείνει στην Ευρώπη μειώνοντας την Ομοσπονδιακή Ευρώπη την οποία εγώ θέλω, τότε εγώ θα επιλέξω να μην έχω μαζί μου το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Η συζήτηση δεν γίνεται μόνο με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το θέμα δεν είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργήσει ο Κάμερον με την εξαγγελία ε, του δημοψηφίσματος. Θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το τίμημα για την Ευρώπη της κατάληξης, της έκβασης. Και μία ερώτηση για να τελειώνουμε. Είναι δυνατόν να συνδυάσει κανείς δύο λύσεις, τις δύο λύσεις. Είναι δυνατόν να υπάρξει ε, μια συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο σε μικρές μεταρρυθμίσεις οι οποίες με πραγματιστικό τρόπο θα βοηθήσουν το Ηνωμένο Βασίλειο ε, να κερδίσει την κυβέρνηση, να κερδίσει ε, είναι συμβατό κάτι τέτοιο με μια Ευρώπη η οποία βγαίνει από την οικονομική κρίση βελτιώνοντας την οικονομική της διακυβέρνηση. Ε, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες ε, έχουν αρνηθεί την είσοδό τους στο ευρώ. πώς μπορούμε εμείς να καταστήσουμε τις μεταρρυθμίσεις μας συμβατές με τα αιτήματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Μικρές μεταρρυθμίσεις, καλύτερη λειτουργία της ρύθμισης, της οικονομικής διακυβέρνησης, περισσότερη επικουρικότητα και ταυτόχρονα να κάνουμε βήματα προς μια πιο ομοσπονδιακή Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που άρχισε η συζήτηση για το τι είδους συμφωνία μπορεί να έχουμε με τον κύριο Κάμερον και φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι μια τέτοιου είδους συμφωνία μπορεί να μην είναι τόσο σημαντική για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ε, ούτως ή άλλως. Η αρχική υπόθεση ήταν ότι χρειαζόμαστε μια συμφωνία για να αποφύγουμε το Brexit. Μετά περάσαμε στο επόμενο στάδιο τι είδους συμφωνία χρειαζόμαστε και τώρα ε, ο Τσάρλς μας είπε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η ιδιαίτερη επιθυμία για αλλαγή για συμφωνία, συγγνώμη, και ο Τσάρλς μας είπε ότι οι μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία της Ένωσης μπορεί να, είναι, να μπορεί να μην είναι επαρκής ε, αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε στο 1975 και δεν, δεν είναι αρκετό αυτό. Κάτι όμως ε, ελπίζουμε ότι θα συμφωνηθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι σημαντικό να υπάρξει ε, μια συμφωνία ε, ώστε να είναι στη σωστή πλευρά του δημοψηφίσματος ο David Cameron και να προσπαθήσουμε βέβαια να κερδίσουμε το δημοψήφισμα. Όμως αν η... Δεν ξέρουμε αν το, το γεγονός ότι θα γίνουν προσαρμογές ε, θα είναι αποφασιστικό για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Η διαφορά που, είχε, που υπήρχε με τη Σκοτία και το δημοψήφισμα τότε δεν ήταν αυτό το οποίο είχε ε, υποσχεθεί στη Σκοτία, αλλά ο λόγος του Γκόρντον Μπράουν, που είχε δείξει τις συνέπειες ε, της αποχώρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο της Σκοτίας και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και οι κίνδυνοι που υπήρχαν. Και και τι θα έχαναν ε, οι Σκοτσέζοι σε αυτή την περίπτωση. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Καλό είναι να έχουμε αυτή τη συμφωνία, ίσως επί ίσονος σημασία ζητημάτων με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά για να κερδίσουμε το δημοψήφισμα μη, επί τη βάση μιας πολιτικής συζήτησης ε, ε, για τις ενδεχόμενες ε, συνέπειες απομόνωσης, για παράδειγμα, του Ηνωμένου Βασιλείου, όχι από οι δομένες από το πρίσμα των ε, μεγάλων επιχειρήσεων, των οικονομικών συνεπειών για τον κόσμο, για τους ε, πολίτες, το ότι δεν θα είναι πια στην ε, ενιαία αγορά, ότι δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε οικονομικές ε, συνθήκες ε, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όπως επίσης ε, και οι πολιτικές συνέπειες μιας απομόνωσης της, του Ηνωμένου Βασιλείου υπάρχει περιθώριο τέτοιου είδους ε, Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε το δημοψήφισμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Φάμπιο. θα ομιλήσω την Ιταλική. Να ευχαριστήσω τους δύο μιλητές για την ενδιαφέρουσα ανάλυση τους και για τα, θέματα που έθεσαν και για την εσωτερική πολιτική και για την ευρωπαϊκή διάσταση και τα θεσμικά συνταγματικά προβλήματα. Θα ξεκινήσω αναφερόμενος σε έναν μεγάλο συνταγματολόγο, Ιταλό τον Τεγκάσπερη, ή μάλλον ε, ένας ε, μέγας πολιτικός, ο οποίος είχε ασχοληθεί με κάποιες εκλογές και αν δω ακριβώς το τι γίνεται σήμερα, βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί πολιτικοί αλλά λίγοι εθνάρχες θα το πω κάπως διαφορετικά, μεγάλοι πολιτικοί. Το θέμα δεν είναι να καταλήξουμε σε μια τακτική απόφαση. Το θέμα δεν είναι να κρίνουμε και να καταδικάσουμε αυτούς που είναι περισσότερο εναντίον της Ευρώπης. Το θέμα είναι να κάνουμε μια σαφέστατα στρατηγική απάντηση στον Κάμερον και στο κόμμα του. Αυτό έχει στρατηγικές συνέπειες βέβαια και οι στρατηγικές συνέπειες είναι και το λεγόμενο ατύχημα στην πορεία, το Brexit, το οποίο δεν θέλει κανείς ακόμα και από αυτούς οι οποίοι προτείνουν το δημοψήφισμα, αλλά συμβαίνει λόγω παραγόντων εξωτερικών όπως ο οικονομικός κύκλος, όπως τα εσωτερικά προβλήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ρητορική κτλ. Ίσως από τη μία έκανε λάθος ο Κάμερον και να ξαναγίνει αυτό το οποίο συνέβη στο δημοψήφισμα στη Σκοτία φοβήθηκαν τις συνέπειες και κατάφερε τελικά να πετύχουν όμως κάποιες παραχωρήσεις οι οποίες θεωρούνται θετικές πολιτικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια νομίζω ότι δεν αντιμετωπίζουμε σωστά την κατάσταση. Ακούω πολλούς να λένε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα τη Βρετανία και πώς να μπορέσει το εκλογικό σώμα στη Βρετανία να κατανοήσει. Να βρούμε στρατη... εκστρατείες στρατηγικής ενημέρωσης κτλ. Όχι, εγώ νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με πιο θαραλέο τρόπο και με πιο λογικό τρόπο. Έλεγα πριν ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μια αναθεώρηση των συνθήκων έχουμε να κάνουμε με ασυμμετρίες οικονομικές και με μια τεράστια οικονομική κρίση η οποία έχει δείξει γυμνές τις αντιφάσεις που μαστίζουν την Ευρώπη και που ήταν συγκεκαλυμμένες στο παρελθόν. Στα πλαίσια αυτής της λογικής λοιπόν μπορούμε να συνδέσουμε την προβληματική μας και με τις διεκδικήσεις κάποιες από αυτές των Βρετανικών αρχών. Την κοινωνική διάσταση, την ενίσχυση του ελέγχου των αρχών θα υπάρξει άλλωστε και μία έκθεση του Φερχόστατ που θα ασχοληθεί με ακριβώς το συγκεκριμένο όραμα το οποίο θα πρέπει να έχει το Κοινοβούλιο γύρω από τα θέματα αυτά. Ε, μήπως λοιπόν αντί να συζητάμε το πώς θα πείσουμε το εκλογικό σώμα να δείξουμε ότι και στις υπόλοιπες χώρες γίνεται μια προσπάθεια η οποία οδηγεί στη μεταρρύθμιση των συνθήκων να πείσουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι ένας μηχανιστικός οργανισμός που υποκύπτει στην οικονομική κρίση, αλλά ένας οργανισμός ζωντανός, ζωηρός που αποτελείται από πολλές χώρες και αυτή η μορφή συνεργασίας δείχνει την ζωτικότητα και την ενέργεια που έχει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και σε ένα-δυο χρόνια θα γίνει μια διακυβερνητική συνάντηση όπου τέτοιου είδους ε, προβλήματα θα αντιμετωπιστούν. Οπότε τότε εφόσον βελτιώσουμε τη λειτουργία της Ένωσης τότε θα κερδίσουμε και τις καρδιές των Βρετανών. Νομίζω ότι μια Ευρώπη που ανανεώνεται είναι μια Ευρώπη η οποία θα πείσει τους διστακτικούς. I'm an MEP. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι από την Ιρλανδία και αν το Brexit συμβεί τότε θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Κάποιοι θα πούνε καλό αντίκτυπο, κάποιοι θα πούνε αρνητικό για την Ιρλανδική οικονομία και γι' αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τη δικιά μου την πατρίδα και είναι καλό που μπήκαμε σε λεπτομέρειες. Ακούω πολλούς να λένε για υπνοβασία προς το Brexit. Όταν το ακούω αυτό, νομίζω ότι η αλαζονία θα μας φέρει στο Brexit, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και τώρα ακούμε τέτοιου είδους διατυπώσεις και ξέρω, Ζαν Κλοντ, ότι δεν προσπαθείς να προσβάλλεις τους Ιρλανδούς με τα σχόλιά σου, αλλά η αλαζονία είναι να απορρίπτει τι απόψει των άλλων ανθρώπων και όταν δεν συμφωνούμε να του λέει απλώ δεν καταλαβαίνει. Όταν η Ιρλανδία ψήφισε όχι στα δύο δημοψηφίματα, μα είπατε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Και αυτό έβλεψε πιο πολύ του ευρωσκεπτικιστέ, γιατί σε κάποιου που έρχονται μια μορφωμένη χώρα δεν του αρέσει να του λένε ότι όταν δεν συμφωνούμε με κάποιου άλλου απλώ δεν καταλαβαίνουν. Έχω τρει κόρε και πολλές φορέ κάνω και εγώ το λάθο να το πω αυτό. Και είναι παιδιά. Και δεν καταλαβαίνω όντω, αλλά και πάλι είναι λάθο. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να φύγει αυτή η αλαζονία. Μπορεί να μην είναι προμελετημένη, αλλά είναι ένα γενές, μια γενή συνήθεια. Να του ρωτήσω, ψήφισαν ναι επειδή δεν κατάλαβαν. Και υπάρχει και αλαζονία όταν ακούω ότι χρειαζόμαστε ε, πίεση στους πολιτικούς ηγέτες, ακόμα και αν δεν πιστεύουν στην περαιτέρω εμβάθυνση του ευρωπαϊκού ε, προγράμματος, ακόμα και αν δεν το πιστεύουν. Επίσης, αλαζονία υπάρχει και δεν μου αρέσει καθόλου ο τύπος, δεν θέλω να εκφραστώ για τον τύπο γιατί θα ακουστώ άσχημα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θέλουν να πουλάνε αντίτυπα και ένας λόγος του ευρωσκεπτικισμού είναι επειδή πολλοί αναγνώστε ευρωσκεπτικιστέ. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα και να ακούσουμε τους πολίτες. Εγώ ήμουνα υπέρ τη Ευρώπη και τώρα έχω γίνει ευρωσκεπτικιστής της αριστερή πτέρυγα κιόλα. Για φανταστείτε, Ένα από τους βασικούς λόγους και αν είσαι από ένα περήφανο έθνος σαν τη Βρετανία, θα το καταλάβετε αυτό όταν λες ναι, για να πας πιο κοντά στην καρδιά της Ευρώπης και πρέπει να λάβεις σοβαρές αποφάσεις, ανοίγεις τον κληπτικό σταθμό και, λέ, και βλέπεις ε, τη Μέρκελ και τον Ολάν να κάνουν ε, ανακοινώσεις. Ακόμα και στο πιο χαμηλό επίπεδο στο δούμε. Αν είχαμε μια επιτροπή με 20 ανθρώπους και έπρεπε να λάβουμε μια σοβαρή απόφαση, αν οι δύο πιο πλούσιοι γείτονε και πιο ισχυροί σωματικά έβγαιναν και έλεγαν αυτή είναι η κανόνε για το κράτος μας, κράτος μας. εμείς θα ηγηθούμε. Τι θα πιστεύατε, άρα αν θέλεις να πρέπει να, αν θέλετε να δουλέψει όλο αυτό πρέπει να φύγετε από αυτήν την οτροπία. Εκατό χρόνια του χρόνου από, είναι πέτυχη της περιφέρεια από μια αυτοκρατορία Πώ θα λειτουργήσει όμω η κοινότητά μα, αν απαξιώνουμε ανθρώπους. Υπάρχει και μια απειλή σε αυτό το διάλογο. Η Μεγάλη δεν είναι κυρίαρχο κράτο. Γιατί πρέπει να του πείσουμε να μείνουν απειλώντα του. Παραδείγματο χάρη ε, θα υπακτρολίουμε τι ε, συμφωνίε με τα συνδικάτα κτλ. Πιστεύω ότι και πολλέ επιχειρήσει δεν θα συμφωνούσαν με το να σταματήσουν τι ε, συνεργασίε με βρετανικέ επιχειρήσει εξαιτία των απόψεών σα. Βλέπω έναν πολύ ενδιαφέρον διάλογο, αλλά το θέλω πιο ευροσκεπτικιστικό το διάλογο. Πολλοί λένε ότι είναι κακή λέξη ο σκεπτικισμός. Πρέπει να τα αμφισβητούμε όλα αυτά που διέπουν τη ζωή μας και να τα αμφισβητούμε όλα. Και όταν είμαστε σκεπτικιστές, δεν είναι κακό. Πρέπει να αρχίσουμε να ρωτάμε, να θέτουμε ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τους ε, ομιλητές μας ε, να σχολιάσουν. Θα αρχίσω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Η πρώτη από την Ισπανίδα κυρία εδώ δεξιά μου, κατά πόσο θα ήταν καταστροφή να υποκύψουμε στο τραγούδι των θηρήνων και στο λαϊκισμό και να υπονομεύσουμε το ευρωπαϊκό σύστημα. Αυτό εξαρτάται για το τι, από, το τι, από το τι πιστεύετε ότι είναι οι συνέπειες ενός Brexit. Κανένας δεν μίλησε για το τι σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα Brexit και ελπίζω ότι κάποια άλλη στιγμή με ε, άλλους παρευρισκομένους θα συζητηθεί αυτό το θέμα. Ε, το, α, το τι απαντάτε σε αυτή την ερώτηση ε, ε, έχει άμεση σχέση με το τι μπορείτε να κάνετε και τι είστε διατεθειμένοι να κάνετε για να παραμείνει η Μεγάλη Βρετανία ε, κατά πόσο δηλαδή υπάρχουν συνέπειες ε, στην εξωτερική πολιτική, στην οικονομία. Ε, αν θεωρείτε ότι είναι τεράστιες ε, οι συνέπειες, ίσως θα έπρεπε να ακούσετε τις ειρήνες και ίσως αν δεν τις ακούσετε και αφήσετε τους Βρετανούς να φύγουν, μπορεί να το μετανιώσετε αργότερα. Δεν λέω ότι μπορεί να είναι καταστροφή για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση αν ε, η Μεγάλη Βρετανία αποχωρήσει, αλλά δεν είμαι και πολύ αντικειμενικός για αυτό το θέμα. Ο Ιταλός ε, συνάδελφος είπε το εξής, υπάρχει πολλές φορές η άποψη ότι η Βρετανία θα έπρεπε να φύγει και να έχει συνθήκες με την Ευρωζώνη και τέτοιου είδους επιχειρήματα. Ε, και ότι πολλοί κόσμος ε, μπορεί να μην θέλει να συγχροτίζεται πια με τους Βρετανούς γιατί η εικόνα των Βρετανών έχει αμαυρωθεί δεν είναι δυνατόν ε, τα πράγματα να οργανώνονται με τόσο απλοϊκούς όρους το να είναι κανείς ή να μην είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλο θέμα και έχει να κάνει και με το θέμα της συμμετοχής στην Ευρωζώνη ή όχι Είχατε γράψει ένα άρθρο στο Sunday Times ε, και είχατε εκφράσει κάποιες επικρίσεις για την Βρετανική κυβέρνηση. Το άρθρο αυτό στο οποίο αναφέρεστε ε, δεν ε, επικρίνει ουσιαστικά ε, τα επιδόματα για τους ε, μετανάστες και δεν επικρίνει την, κυκλοφορία της, ε, την ελευθερία της κυκλοφορίας και την ελευθερία του εργάζεσθε στις, στα διάφο, στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ένας φίλος από την Ισπανία ρώτησε το εξής, θα έπρεπε το φεντεραλισμό να τον ε, αφήσουμε στην άκρη αν ε, δεχθούμε τις διεκδικήσεις της Βρετανικές. Εγώ δεν νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ε, της Ευρώπης είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι χώρες που γνωρίζω εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο και που τις γνωρίζω καλά είναι η Γαλλία και η Γερμανία και όταν μιλάω στους πολιτικούς τους μας λένε ότι έχουν ενδιασμούς για το να θέσουν μια, ένα δημοψήφισμα στις χώρες τους για την εκχώρηση περισσότερων εξουσιών στις ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότερες χώρες δεν θέλουν ή τουλάχιστον έχουν ενδιασμούς στην εκχώρηση αυτή. Οπότε αν το υπονοείτε κάνετε λάθος. Δεν είναι... Αν, ακόμη και αν φύγουν οι Βρετανοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα υπάρξει ομόσπονδη η Ευρώπη, τουλάχιστον όχι σύντομα. Το να γίνουν ε, υποχωρήσεις προς την ε, ε, Βρετανία δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα καθυστερήσει μια ομοσπονδία ευρωπαϊκών κρατών. Ουσιαστικά η άποψη των Βρετανών της, του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου είναι ότι πρέπει περισσότερο να ενσωματωθεί η Μεγάλη Βρετανία. Ας πούμε τα ευρωομόλογα μας αρέσουν πολύ. Δεν σημαίνει υποχρεωτικά δηλαδή ότι εμείς θέλουμε να ε, διαλέγουμε και να παίρνουμε. Και τέλος, αν θα μπορέσει να υπάρξει ένας λόγος τύπου Gordon Brown, α, μάλλον πριν πάω εκεί, είχατε πει εσείς ότι οποιαδήποτε συμφωνία ε, δεν θα επηρεάσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο. Είναι γεγονός ότι το θέμα θα είναι τα υπέρ και τα κατά του εντός και εκτός της Ένωσης. Αν ο Κάμερον μπορεί να καταλήξει σε μια αρκετά πιστική συμφωνία, τότε ένα τμήμα του κόμματός του θα μετακινηθεί και το θα τον υποστηρίξει. Και αυτό θα επηρεάσει και τις πολιτικές συζητήσεις αλλού. Είναι σημαντικό λοιπόν το τι θα καταφέρει να επιτύχει ο Κάμερον. Ορισμένα ζητήματα βέβαια της εκστρατείας θα, θα έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι άλλα. Αυτό που είπατε για το λόγο του Γκόρντον Μπράουν, ε, αν ο Τζον ε, ε είπε ότι ε, ναι, καλύτερα θα ήταν να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, κοιτάξτε, τώρα ε, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδου παραλληλισμούς για λόγους που δεν μπορώ να ε, εμβαθύνω αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν επιχειρήματα για υπέρ του παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βρετανία είναι εσωστρεφή εσωστρεφής χώρα, ε, πολύ εσωστρεφής, ε, ε, θέλει να παραμείνει έτσι ή θέλει να χαρακτηριστεί από μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Αυτό είναι το επιχείρημα ε, το οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε ίσως την τελευταία στιγμή. Η ανάγκη τώρα της ε, διαπραγμάτευσης ε, των εμπορικών συμφωνιών, αυτό δεν προκύπτει από την υπεροψία κανενός. Αυτό προκύπτει από την νομοθεσία. Αν έχει κάποιο υπογράψει μια συμφωνία και μετά αποχωρεί από τον οργανισμό που την ε, συνήψε, πρέπει να την ε, διαπραγματευτεί εκ νέου. Ναι, απλώς δεν πρέπει να, είμαστε, ε, να μην είμαστε ρεαλιστές. Είναι αμφίδρομο το εμπόριο θα ήθελα πάρα πολύ να δω ε, τι θα γίνει με τους δασμούς. Ε, ε, είναι προς όφελος και των δύο πλευρών να συνεχιστεί ένα εμπόριο και απλώς εκφοβισμός είναι αυτό, δεν χαζός ο κόσμος. Βλέπουν μέσα από αυτά τα εκφοβιστικά επιχειρήματα. Ναι, λέει η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο ομιλητές. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν για την παρουσία σας. Δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να κάνουμε τέτοιου είδους ε, συζήτηση. Θα υπάρξουν και άλλες συζητήσεις στο μέλλον. Μπορούμε επίσης να φανταστούμε ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ δύσκολοι για τον κύριο Κάμερον, γιατί υποθέτω ότι οι επιθέσεις ε, γίνονται όλο και ε, εντονότερες και υποθέτω ότι χρειάζεται υπευθυνότητα και από τη δική μας πλευρά να μην ρίξουμε λάδι στη φωτιά. Νομίζω ότι όλα αυτά που ακούστηκαν σήμερα και είχαμε και την ευκαιρία να εκφράσουμε τις απόψεις ήταν πάρα πολύ χρήσιμα για όλους. Θα συνεχίσουμε ε, τον προβληματισμό μας και ας ελπίσουμε ότι η μεγάλη Ευρώπη θα επιβιώσει. Θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτό το σημείο τη ημερήσιας διάταξη. Όμω παρακαλώ να παραμείνετε γιατί έχουμε και άλλα σημεία στην ημερήσια διάταξη. Δεν έχουμε ολοκληρώσει τη συνεδρία. Ευχαριστώ. Um, Ο Ράινερ Βίλαντ είναι εδώ, οπότε μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξής μας, ε, που είναι η έκθεση της ομάδας εργασίας ε, υπό την προεδρία του κυρίου Βίλαντ από τον Ιανουάριο εργάζεται αυτή η ομάδα για την αναθεώρηση των, του εσωτερικού κανονισμού. Ράινερ, είσαι έτοιμος να μας κάνεις την παρουσίασή σου, έχεις το λόγο. Μισό λεπτό να βάλω τα γυαλιά μου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας δώσω αυτή την διάμεση έκθεση η οποία δεν είναι απλή όπως θα καταλάβετε διαβάζοντάς την αυτή η Επιτροπή Είχε μια σύσταση από τους συντονιστές 7 Οκτωβρίου του 2017 ε, να δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας για να προγραμματίσει μια αναθεωρημένη μερικιά διάταξη. Συμφωνήθηκε αυτή η ομάδα στις 6 Νοεμβρίου και ανήκουν άτομα και από το ΕΛΚ και άλλοι συνάδελφοι που εκπροσωπούν τις υπόλοιπες ομάδες, ο Κόρμπιτ, ο Γιατσόφσκι, ο Ντεγκέρινγκς, ο Σούλτς, η Αντινόλφη, ο Άντερσον και ο Άνιμανς. ο οποίος έχει αλλάξει στάτους, αλλά αρχικά ήταν μέλος, τώρα επιβλέπει... Noch mit. Äh, wir haben einen, Για τους μη εγγεγραμμένους είναι επόπτης. Και τώρα θα τα διαβάσω στα αγγλικά να εντοπίσουμε ενδεχόμενα λάθη, ασυνέπειες, καθώς και διατάξεις που είναι πλέον απαρχαιωμένες και χρειάζονται προσαρμογή εξαιτίας των εμπειριών των τελευταίων χρόνων. Είναι πολύ ξεκάθαρη η εντολή, όπως βλέπετε. 13 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο είχαμε την πρώτη συνεδρίαση και εγώ επιλέχθηκα ως ε, πρόεδρος. Ακόμα και δεν υπήρξε επίσημη απόφαση κάναμε την κατανομή και εγώ έγινα πρόεδρος, ο Κόρμπιτ ε, έγινε εισηγητής. Βλέπετε ότι έχουμε ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα και εξακολουθούμε να το έχουμε από το 2012. Οργανώσαμε συναντήσεις, η τελευταία ήταν 9 Ιουλίου πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα. Έχουμε κάθε μήνα δύο συνεδριάσεις και τώρα θα παρουσιάσουμε ήδη ένα αποτέλεσμα. Ο στόχος είναι φιλόδοξος και το έχουμε καταλάβει πλέον και δεν θα μπορέσουμε ε, να ολοκληρώσουμε αυτά που θέλαμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Είχαμε ανταλλαγή απόψε στη τελευταία συνάντηση που αφορούσε το, τα First Reading Agreements Είχαμε δύο έμπειρους συναδέλφους, τον κύριο Σφάβ και τον Άικαουτ. Η επόμενη συνεδρία είναι στις 10 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο. Επιπλέον, δημιουργήσαμε μια ομάδα διοικητική για το πρόγραμμα αυτό που υποστηρίζει την ομάδα εργασίας από δύο πλευρές. πρώτα θα προσπαθήσει να εντοπίσει τα προβληματικά σημεία στα κείμενα ε, και να τα επισημάνει στην ομάδα εργασίας και περιορίζεται αυστηρά σε πράγματα που δεν έχουν ουσιαστική πολιτική αξία. Κάτι που αφήσετε λοιπόν σημειώνεται και παράλληλα κάνει και προτάσεις αυτή η ομάδα Επίσης έχουμε το σύστημα στα εργασία, να θέτουμε ανοιχτά ερωτήματα και να τα συζητάμε και να αποφασίζουμε πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση και μετά ζητάμε από την ε, ομάδα αυτή, την προγραμματική ομάδα να μας κάνει προτάσεις και τη διατύπωση να δούμε αν υπάρχουν ε, αντικρουόμενα στοιχεία, ώστε να καταλήξουμε στη σωστή διατύπωση επίσης και να συζητήσουμε τις προτάσεις αυτές περαιτέρω. Äh, Έχουμε ολοκληρώσει το 1 τρίτο του τίτλου 1 που αφορά ε, τα μέλη και τις ομάδες. Στο δεύτερο τίτλο έχουμε την ομοθεσία, τον τριπολογισμό και άλλες διαδικασίες. θα είναι κάπως δύσκολο γιατί η θέση μου είναι διφορούμενη υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα, όπως είπαμε και νωρίτερα, ως προς τον κανονισμό, αντικρώμενα συμφέροντα μεταξύ των ομάδων. Στις πολιτικές ομάδες γίνονται συζητήσεις και για μονομένα ερωτήματα ή θα προκύψουν ερωτήματα ενδεχομένως. Και παρακαλώ πάντως τους προσώπους των πολιτικών ομάδων να συζητήσουν τα θέματα αυτά στο πλαίσιο των ομάδων τους. Δεν θέλω να εμβαθύνω στο θέμα, αλλά υπάρχουν ήδη κάποια ερωτήματα που θύχτηκαν και που φάνηκε ότι ε, δεν λαμβάνουν χώρα αυτές τις συζητήσεις στις ε, πολιτικές ομάδες. Κάνω επισημάνσεις ε, γυρνώνω συναδέλφους, ε, κάποιους κοντινούς μου, δεν το κρύβουν καπνιστής και στο καπνιστήριο συναντώ πολλούς από άλλες εθνικότητες, άλλες ε, πολιτικές ομάδες. Και εκεί πέρα γίνονται φυσικά συζητήσεις. Και τελικά συμφωνήσαμε ότι δεν θα κάνουμε συνεδριάσεις κυκλοφορών των θύρων, και ότι μετά από κάθε συνεδρίαση θα γίνονται συνεδεύξεις τύπου, μετά για ενημέρωση και δεν θα γίνονται αυτές οι συνεδεύξεις πρωτού υπάρξει πρώτα συμφωνία. Να κατονομάσω και κάποια άλλα θέματα τα οποία μας απασχολούν και για τα οποία συζητάμε. Όπως είπα, Πρέπει να βελτιώσουμε τις διαδικασίες εντός των πολιτικών ομάδων. Είμαστε στον τίτλο 1, όπως είπα. Ακόμα. Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει. Θέματα ασυλίας Έχουμε συζητήσει. Υπάρχουν όμως και άλλα ανοιχτά ερωτήματα. Όπως τον τους χάρη. Πώς θα γίνονται οι εκλογές. Και... betreffend die στο Κοινοβούλιο για τις αρμοδιότητες του Προέδρου, του Προεδρίου, των κοσμητόρων και οι κανόνες για το σχηματισμό των πολιτικών ομάδων, με ποιες νομικές συνέπειες και πώς αυτές οι ομάδες θα διαλύονται και πάλι με ποιες επιδράσεις. Πάμε μετά στο δεύτερο τίτλο. όπου βρήκαμε κάποιες διατυπώσεις που αφορούν γενικές ρυθμίσεις νομοθετικές, αλλά υπάρχουν και σχετικές διαδικασίες στις επιτροπές που χρειάζονται και αυτές, επειδή έχουν και αυτή η συζήτηση, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι εκθέσεων. Επίσης υπάρχει και το θέμα των γνωμοδοτήσεων ποια θα είναι η ταχύτητα επεξεργασίας τους και να πω σε αυτό το σημείο ότι 12-14 άτομα σε μια επιτροπή προσπαθούν ε, γρήγορα να ολοκληρώσουν ε, τη δουλειά τους να ολοκληρώσουν ε, τη γνωμοδότηση και έτσι κανείς δεν... και μετά καταλήγουν μετά από αυτή τη βιασύνη να μην λαμβάνει και κανείς υπόψη αυτή τη γνωμοδότηση. Επίσης, η συνεργασία των επιτροπών. Πώς θα ξεδιπλώνεται αυτή η συνεργασία. Είδαμε τον συνάδελφο Άικαουτ και τον ε, συνάδελφο Σβάμπ. για να συζητήσουμε για τις νομοθετικές διαδικασίες, για τους τριμερείς διαλόγους και τις συμφωνίες για το εμπόριο, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να πάρει την εντολή, να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με διαφάνεια. που θα είναι εξασφαλισμένη στη διαφάνεια, χωρίς όμως να υπάρχει παράλληλα ο κίνδυνος ε, να χαθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα. Άλλο θέμα είναι το πόσο συχνές είναι οι εκθέσεις πρωτοβουλίας. Στην τελευταία νομοθετική περίοδο ήταν πολύ συχνές οι εκθέσεις πρωτοβουλίας και είχαμε την αίσθηση ότι αυτό δεν ε, είχε αποδοχή Επίσης το first reading, η πρώτη ανάγνωση είναι ένα θέμα που μένει ανοιχτό. Δεν ξέρω αν συζητηθήκε σε όλες τις ομάδες. Έκανα πρόταση να ξεκινήσει ο διάλογος künftig den Kommissionspräsidenten in offener Abstimmung wählen. Να αποφασίσουν για τον τρόπο ψηφοφορίας, να μην υπάρχει μυστική ψηφοφορία, να υπάρχει συνέπεια, να υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία. Και υπάρχει και ένα άλλο σημείο στο οποίο θέλω να πιστήσω την προσοχή σας στην προηγούμενη Βουλή δεν ήταν τόσο έντονο αυτό το θέμα, αλλά τώρα πλέον υπάρχει ένα mail που κυκλοφορεί όπου δεχόμαστε συγχαρητήρια για την εκλογή μας και ουσιαστικά Υπάρχει ουσιαστικά ένας συναγωνισμός για τον ποιον θα έχει πιο πολλές ε, ε, παρεμβάσεις, ποιος παίρνει πιο συχνά το λόγο, ποιος κάνει τις πιο πολλές προτάσεις τροπολογίας, γραπτά ερωτήματα προς την Επιτροπή. Λοιπόν, σε αυτή την κλίμακα, στην κατάταξη, βρέθηκα κάπου ψηλά και κατάλαβα ότι είχα πολλές φορές πάρει το λόγο στην Ολομέλεια. Αν και από ό,τι θυμόμουν δεν είχα μιλήσει ποτέ ουσιαστικά σε αυτήν την ομοθετική περίοδο. Απλώς ήμουν συντονιστής, έλεγα ποιος θα πάρει το λόγο ε, μετά, ποιος πριν, αλλά και αυτά θεωρούνται ως ε, παρεμβάσεις. Υπάρχουν πολλά παράδοξα σε αυτή την κατάταξη. Και κάποιο άλλο συνάδελφο που είχε αρρωστήσει είχε πάρει πολύ άσχημη θέση στην κατάταξη. Και τώρα ξαφνικά όλοι ξυπνάνε και λένε οι περισσότεροι ότι δεν είναι σωστή αυτή η προσέγγιση. Είναι μια πολύ σοβαρή λάθος θα έλεγα εξέλιξη. Θα πρέπει μάλλον να μιλήσουμε για τα δεδομένα και τα νούμερα που δίνει προς τα έξω, που διαθέτει το Κοινοβούλιο. Είναι πραγματικά σωστό το, το κοινοβούλιο να λέει ότι υπάρχουν ότι υπάρχουν 37 παρεμβάσεις αυτού του βουλευτή και πρέπει αυτό το, την πληροφορία να τη μεταδώσουμε. Αυτό που ενδιαφέρεται πραγματικά για κάτι τέτοιο μπορεί να το ψάξει μόνο του, αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε αυτή την ποσοτική προσέγγιση στο θέμα. Αυτό δεν αφορά τον κανονισμό. Όμως υπάρχουν πολλές λάθος εξελίξεις γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που προτιμούν τις στατιστικές και όχι την πολιτική. Προτιμούν να κάνουν στατιστικές παρά πολιτική. Είχαμε πολλέ ψηφορίες στην προηγούμενη ε, θητεία. Πολλέ προτάσεις μάλλον ε, και πολλές από αυτές ε, τις πέβαλαν γραπτός. Πάνω από 70.000 υπήρξαν. Πολλές ήταν και αποτέλεσμα copy-paste, χωρίς νόημα, μόνο για να καταμετρηθούν, γι' αυτό το λόγο και μόνο. Επίσης, τα ερωτήματα στην Επιτροπή. Και εκεί είχαμε έναν τεράστιο αριθμό και ρωτήθηκε προηγουμένως αν η Επιτροπή είχε γνώση της θνησιμότητας των βρεφών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί μάλλον τα ξεχωριστά τη Γερμανία κτλ. 28 ξεχωριστά ερωτήματα και σήμερα ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα, ότι δεν πρέπει να κάνουμε πάνω από πέντε, να υποβάλουμε πάνω από πέντε ερωτήσεις. Και λέω τώρα ότι αν αφαιρέσουμε αυτή την ποσοτική προσέγγιση, τότε πολύ γρήγορα θα ομαλοποιηθούν αυτά τα νούμερα και θεωρώ ότι αυτοί οι βουλευτές που θέλουν για πολιτικούς λόγους ε, να θέσουν ερωτήματα δεν θα πρέπει να περιορίζονται στην πράξη. Μίλησα με τη συνάδελφο και είπα ότι χρειαζόμαστε επιγόντως τις αλλαγές αυτές μέχρι 1η Ιανουαρίου ώστε να έχουμε τα πρώτα στατιστικά αποτελέσματα και να ρωτήσουμε να δούμε μάλλον αν όντως αυτή η προσέγγιση, αυτή η ενέργεια είναι χρήσιμη για τις εργασίες του Κοινοβουλίου ή αν μέσω της ομαλοποίησης αυτής που ανέφερα πριν θα έχουμε πιο καλά αποτελέσματα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σημείο αυτό και προσωπικά θεωρώ ότι κανείς στην ομάδα εργασίας πιστεύω ότι κανείς δεν θέλει να περιορίσει τα προσωπικά, ε, τα δικαιώματα που έχουν οι ευρωβουλευτές. Κανείς δεν έχει αυτή την πρόθεση. Και αυτό που θα ήθελα είναι να έχουμε πιο λογικές και λιγότερες ερωτήσεις προς την Επιτροπή, ώστε να πει και η Επιτροπή ότι έχετε λιγότερες ερωτήσεις, μας υποβάλλετε λιγότερες ερωτήσεις, αλλά τώρα μπορούμε, να, να σας απαντήσουμε με πιο ε, λογικό τρόπο. Λοιπόν, το δεύτερο εξάμεινο συνεχίσαμε αυτό το... Ασχοληθήκαμε και συνέχεια με αυτό το θέμα. Οποιοςδήποτε έχει απορίες ε, να έρχεται και να μας ε, ζητάει πληροφορίες. Παρακαλώ και τα μέλη ε, τα μέλη της ομα, των ομάδων να δώσουν και αυτά να, να προετοιμάσουν μια ενδιάμεση μελέτη ώστε να έχουμε ένα συνολικό αποτέλεσμα που θα το συζητήσουμε και θα το εντάξουμε στις εργασίες της ε, ομάδας εργασίας μας. Θα ήθελα να έχουμε και έναν ε, εισηγητή. Θεωρώ ότι πιο κατάλληλος είναι ο κύριος Κόρμπετ που έχει ασχοληθεί προηγουμένως και πιο εντατικά με τον ιστορικό κανονισμό και πιστεύω ότι θα εμπλουτίσει το έργο της ε, Επιτροπής μας. και να μπορέσουμε στη συνέχεια να εφαρμόσουμε στην πράξη τα αποτελέσματα και στα μήτερ του 2017 ε, ε, ανάμεσα ε, στα μισά του 2007 να τεθούν όλα αυτά σε ισχύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στο Κόμπετ. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Ο κ. Βιλάντερ μας έδωσε μια σωστή περιγραφή για το που είμαστε. Προεδρεύει της ομάδας εργασίας με πολλή ικανότητα και μας διευθύνει σωστά. Υπάρχει μια πολύ καλή ατμόσφαιρα σε αυτήν την ομάδα εργασίας. Πριν ξεκινήσουμε υπήρχαν φόβοι ότι θα υπήρχαν συγκρούσεις ανάμεσα στις μεγάλες ομάδες και τις μικρές ανάμεσα στους δεξιούς και τους αριστερούς. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ επικοδομητική η κατάσταση. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα έτσι ώστε το κοινοβούλιο αυτό να δουλέψει καλύτερα. Νομίζω λοιπόν ότι θα συνεχιστεί προς την κατεύθυνση αυτή όταν έχουμε σοβαρές διαφορές για κάποια συγκεκριμένα θέματα, α και είναι τεχνικά τα περισσότερα, οι διαφορές δεν αφορούν ομάδες μεταξύ τους, αλλά το εσωτερικό των ομάδων. Ο κύριος Βίλαντ έδωσε το παράδειγμα ε, της ψηφοφορίας ε, για τον πρόεδρο της Επιτροπής. Θα πρέπει να είναι κρυφή ψηφοφορία ή ανοιχτή. Κάποιοι θεωρούν ότι η μυστική ψηφοφορία προστατεύει το Κοινοβούλιο από την πίεση των κυβερνήσεων γιατί στο παλιό σύστημα επέλεγαν τον πρόεδρο της Επιτροπής και καλούσαν από εμά να τον εγκρίνουμε. Και μας πίεζαν. Τώρα με τον Spitzen Kandidat με το νέο σύστημα όπου ο πρόεδρος της Επιτροπής στην ουσία επιλέγεται ε, μετά τα αποτελέσματα των εκλογών, τα θέματα αλλάζουν. Πολλοί βέβαια ψηφίζουν ε, τα κόμματα τους ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο υποψήφιος πρόεδρος. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ μας, αλλά οι απόψεις των μελών φαίνεται ότι εξαρτώνται περισσότερο από τις παραδόσεις της χώρας από την οποία προέρχονται. Σε ορισμένες χώρες τα κοινοβούλια επιλέγουν τον Πρωθυπουργό ή τον Πρόεδρο, σε άλλες χώρες αυτό δεν γίνεται. Ε, θεωρείται ότι θα πρέπει να γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Σε κάποιες άλλες χώρες η μυστική ψηφοφορία θεωρείται απαράδεκτη. Θα πρέπει ο πολίτης να βλέπει ε, πώς ε, ψηφίζει ο κάθε βουλευτής. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν εντελώς διαφορετικές παραδόσεις. Πάντως, οι διαφορές όπως είπα δεν είναι ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες η μία με την άλλη, αλλά στο εσωτερικό τους. Ήταν εξαιρετική και πλήρης η παρουσίαση του κ. Βίλαντ. Λοιπόν, αυτά δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Α, ο, ο, ο Σόπλιν. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο σε αγνοώ συνέχεια. Σύντομα θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Βίλαντ και τον Κόρμπετ για τη δουλειά την οποία κάνουν. Το θέμα το οποίο θέλω να θέσω είναι αυτό το οποίο απασχολεί γενικότερα σήμερα την Επιτροπή μας. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι στην ουσία ένα πληθωριστικό φαινόμενο. Οδηγεί τον κόσμο προς μια κατεύθυνση η οποία δεν έχει σχέση με την πραγματική δουλειά του Κοινοβουλίου, αλλά ικανοποιεί κάποιες μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ικανοποιεί τις χώρες ε, τις χώρες, τα μέσα ενημέρωσης της χώρες από τις οποίες προέρχεται ο υποψήφιος και η πραγματική δουλειά, ο τρόπος εκπροσώπησης θα έλεγα, ε, η δουλειά την οποία κάνουμε γιατί δυστυχώς οι στατιστικές δεν δείχνουν ε, το τι έχει πολιτικά σημασία. Δεν ξέρω τώρα με ποιο τρόπο και δεν ξέρω σε ποιο φόρουμ το σύστημα αυτό θα πρέπει να μετατραπεί σε ποιοτικότερο. Κάποιες προτάσεις και γενικές σκέψεις έχουν υπάρξει, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα αυτή ε, ε, τη στιγμή λειτουργεί δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικό. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν 17.000 επεξηγήσεις ψήφου, ε, πραγματικά είναι ανόητο αυτό, στατιστικά δεν σημαίνει τίποτα κάθε μέλος θα μπορεί να ζητάει κάθε φορά ε, ε, η παρέμβασή μου να μαγνητοφωνηθεί. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι έχει πάρει το λόγο. Εν πάση Είναι γελία αυτά τα πράγματα, αυτό γελιοποιούμεθα. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα πληθωριστικό φαινόμενο που πρέπει να αντιμετωπιστεί πλέον. Α, Υπάρχει. Μέσα σε όλα δεν βλέπω. Ο κύριος Σόλτς. Η παρατήρηση του κυρίου Σόπλιν με κάνει να θέλω να κάνω και εγώ μία παρατήρηση, γιατί το θέμα είναι πολιτικό. Συζητήσαμε το θέμα της Μεγάλης Βρετανίας σήμερα. τίθεται το θέμα της επεξήγησης ψήφου όταν θέλω να δώσω ακριβώς τους λόγους για τους οποίους αντιμετώπισα μία ψηφοφορία με ένα συγκεκριμένο λόγο. Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν ταυτίζομαι με την πλειοψηφία, δεν ταυτίζομαι με την πολιτική μου ομάδα ίσως και πρέπει να διευκρινιστεί εδώ ότι όταν εμείς εξετάζουμε το θέμα του κανονισμού Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου και έτσι να επηρεάσουμε σωστότερα την πολιτική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν ότι η επεξήγηση ψήφου είναι ένα μέσο το οποίο δεν θα πρέπει να αγνοούμε. Όμως δεν θα πρέπει το μέσο αυτό να γίνει μια απλή στατιστική μέθοδος σόρευσης αναφορών για τον βουλευτή σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Ανησυχώ. Making the decision on the working group, we made it sure that every political group... Κάθε πολιτική ομάδα θα πρέπει να μπορεί να εκπροσωπείται στην ομάδα αυτή. Όταν προετοιμάζαμε την ψηφοφορία για το άρθρο 191 και 101, φάνηκε ότι η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας εργασίας δεν επικοινωνούν σωστά με τις πολιτικές ομάδες. Και πολλοί συντονιστές εξεπλάγησαν από τις ερμηνείες που είχαν δοθεί. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη της ομάδας εργασίας δεν επικοινωνούν σωστά με τις πολιτικές τους ομάδες. Μιλάω για το επίπεδο της ε, Επιτροπής μας, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ανακαλύπτει κανείς ότι οι πολιτικές ομάδες μερικές φορές δεν είναι ιδιαίτερα ευτυχείς από τις προτάσεις οι οποίες μπορεί να προέλθουν από τις συγκεκριμένου τύπου ομάδες εργασίας και που προκαλούν και χιλιάδες τροπολογιών όταν ε, ψηφίζονται. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορεί κανείς ε, να σου ζητήσει Ράιμερ ε, να εξηγήσουμε στις πολιτικές ομάδες όχι μόνο να συνεισφέρουν στην έκθεση αλλά να πούμε στα μέλη μάλλον να επικοινωνούν με τις πολιτικές τους ομάδες για να μην εκπλήσονται οι πολιτικές ομάδες. και να γνωρίζει η Ολομέλεια ότι κάθε τροπολογία θα ψηφιστεί αθεαθής. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε στη φάση αυτή για να επικοινωνήσουμε καλύτερα, να εμπλέξουμε καλύτερα τους συναδέλφους για να υποστηρίξουν τις προτάσεις μας. Δεν ξέρω αν μπορούμε τώρα να κάνουμε κάτι περισσότερο σε σχέση με αυτό το οποίο έχετε ήδη κάνει να επικοινωνήσει κανείς με τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές επιτροπές ή με και τα υπόλοιπα μέλη του Κοινοβουλίου για συγκεκριμένα θέματα. Εν πάση να γίνει η δουλειά μας πιο ανοιχτή και να μην εκπλήσονται από το περιεχόμενο των προτάσεων γιατί μπορεί ίσως τα πράγματα στην παρούσα φάση να μην είναι πάρα πολύ ελκυστικά, να μην είναι πολύ σεξι λέει η πρόεδρος, αλλά στο τέλος της διαδικασίας νομίζω ότι οι προτάσεις της συγκεκριμένη ομάδας εργασίας είναι σημαντικότατες. Και αν ενημερώνουμε σωστά μειώνουμε και τον κίνδυνο απόρριψης, άρνησης της πλειοψηφίας. Ευχαριστώ. Στην πράξη είναι αυτό πολύ σημαντικό Γνωρίζω πώς γίνονται τα πράγματα. Στο πρεδρείο της ομάδες μου ήταν πολλές φορές την διάταξη το θέμα αυτό, αλλά υπήρχαν ε, άλλα πιο σημαντικά πράγματα και ποτέ δεν βρίσκαμε τελικά χρόνο. Το παρουσίασα και στις εθνικές αντιπροσωπείες. Ήμουνα στην διάσκεψη των Πρόεδρων των Επιτροπών. Μίλησα με όλους. όλοι μπορούν να αναφερθούν σε αυτό το θέμα στις ε, ομάδες, στις ομάδες τους και υπάρχουν πάντα ευκαιρίες. Κάνω ό,τι μπορώ ώστε παρά από αυτόν τον τρόπο εργασίας που περιέγραψα να μπορεί οποιοδήποτε να γνωρίζει ακριβώς τι συμβαίνει μέσα στη, στα πλαίσια της ομάδας εργασίας. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια ε, συμπροεδρία στην ομάδα εργασίας και μια εισήγηση από κοινού, να έχουμε συνεισηγητές και στο τέλος να έχουμε έτοιμο το πακέτο και να ήμουν μετά εγώ έτοιμος και στη συνέχεια να έβαζα τον Σάρφο Κόρμπετ να τον έσπρωχνα στη γωνία. Θα μπορούσα να το κάνω και έτσι, αλλά δεν θα ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν θέλουμε να εισηγηθεί το θέμα ως υποσημείωση στην ε, ημερήσια διάταξη, αλλά να αποτελέσει θέμα συζήτηση. I have, uh, Ήμουν εισηγητής για γενικές ε, αναθεωρήσεις του εσωτερικού κανονισμού και όχι στο πλαίσιο μιας επίσημης ομάδας εργασίας και είναι αλήθεια ότι αναπόφευκτα θα υπάρξουν κάποια θέματα που δεν θα υπάρχει συνένεση. Κρίνοντας όμως από το έργο μας μέχρι τώρα το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερος όγκος ε, της δουλειάς μας θα ε, πετύχει συνένεση γιατί ουσιαστικά διαγράφουμε κάποιες, ε, κάποια σημεία που είναι περιτά θα έλεγα. Σίγουρα θα προκύψουν κάποια θέματα, αυτό που ανέφερα πριν και θα υπάρξουν και διαφορετικές απόψεις. Όμως μετά η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα δείξει. Πρέπει να έχουμε κατά για να αλλάξουμε, τον ε, κανονισμό, όπως ένα υψηλό ε, όριο πλειοψηφίας. Δεν θέλουμε μια οριακή πλειοψηφία, θέλουμε μια ε, συμφωνία που θα χαίρει ευρείας αποδοχής. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θέλω να σας ευχαριστήσω για την δουλειά σας. Όχι, δεν είναι το τελευταίο σημείο στην ημερησία διάταξη. Απλώ αναφέρομαι στη συγκεκριμένη ομάδα εργασία. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Θέλω να σα ενημερώσω και αυτά που αποφάσισαν οι συντονιστέ σήμερα. Αποφάσισα ότι το ΕΛΚ θα αναλάβει την ε, εφαρμοστική έκθεση για τη σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια το ECR θα αναλάβει την έκθεση για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα έκθεση Τριτροπής του 2014 και αποφασίσαμε να μην ε, κάνουμε άλλες προτάσεις ε, για ψηφίσματα. Όσον αφορά τις αποστολές, αποφασίσαμε η αποστολή στο Λονδίνο να λάβει χώρα στις 16-17 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Αποφασίσαμε να την ε, ακυρώσουμε γιατί ε, συνέπιπτε με την επίσκεψη στην ε, Washington. Θα αποφασίσουμε στην επόμενη συνεδρία των τονιστών για την επίσκεψη στην Αθήνα και επίσης ανέγκριναν τις συνεδριάσεις της ΑΦΚΟ για το 2016. Δεν υπάρχουν αντίθετε απόψει και θεωρώ ότι εγκρίνονται από την Επιτροπή και να σας ενημερώσω επίσης ότι έχουμε την επόμενη συνεδρίαση Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου το απόγευμα και 22 Σεπτεμβρίου την Τρίτη το πρωί. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχει λήξει η συνεδρίαση.